Συνάδελφοι, καθίστε να ξεκινήσουμε τις σημερινές εργασίες ε, με την ψηφοφορία επί της έκθεσης Taylor για τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου πείτε ποιος δεν έχει την κάρτα μαζί του για να ψηφίσει κύριος Κράμερο, ο κύριος Αλχαντραουή θα πρέπει να μας λέτε λοιπόν τι ψηφίζετε κάθε φορά. Λοιπόν, κάνουμε μία επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ντέμπορα, ψήφισες κι εσύ. Πάτησες το κουμπάκι. Μάλιστα. Όλοι εντάξει. Ωραία. Δεν έχουμε ζαβολιές. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Έκθεση Taylor για τα δικαιώματα αεροπορικών επιβατών, παράγραφος 1, ΙΜΚΟ 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Κατόπιν 16, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Οπότε 15 καταπίπτει. 17 υπέρ. Κατά. εποχέ. Δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Συν ένα συν και ένα πλήν. Το ΕΛΚΑ έχει έναν παραπάνω. Μάλιστα. Πέρας. Και απορρίπτεται. 21 κατά. Ήμκο 2 και 4. Μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική α με χωριστή ψηφοφορία που ζήτησαν οι συντηρητικοί οπότε σε δύο μέρη μέρος πρώτον θεωρεί μέχρι και τις λέξεις Ευρώπη στην Ευρώπη και δεύτερο μέρος από το δέρφο πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά αποχές δεκτό. Οπότε πάμε σε βαστική β. Υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 33 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική C με προφορική τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών. Αντιρρήσει για την προφορική τροπολογία. Όχι. Με την προφορική τροπολογία λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 Μαρινέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική D. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49. Γκρίσμπεκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την επαληθεύσουμε. 49. Νομίζω πως έχει υιοθετηθεί, αλλά άρχεται η ψηφοφορία. voted. Ψήφισαν όλοι. Ναι, συν 2 υπέρ. Πέρας. Δεκτή. 28 με 16. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή και σας ευχαριστώ. 51 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 51 άρχεται η ψηφοφορία συν 2 υπέρ ψήφισαν όλοι πέρας 22 υπέρ 21 κατά δεκτή να είναι δύο που δεν έχουν κάρτα ψηφοφορίας Άρα γίνεται δεκτή. Το συμφωνήσαμε στην αρχή, το δεχτήκατε. 48 σενάλοβα. Καταπίπτει. Και περνάμε στην 52. Αγιάλα Σέντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα την επαληθεύσουμε. Την 52 της κυρίας Αγιάλα Σέντερ. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Μάικλ. Συν δύο υπέρ. Οπότε γίνεται δεκτή. Συμβαστική ή. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 φώστερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 Βότμαν Κόλ υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 70 νομίζω πως έγινε δεκτή άρχεται η ψηφοφορία ε, δείξτε μας τότε κάντε ένα νόημα Μάικλ μάλιστα δύο υπέρ και μία ψήφος κατά επιπλέον πέρας της ψηφοφορίας 31 με 13 δεκτή Ήμκο 18 καταπίπτει. 67 υπέρ. Όχι, συγγνώμη. 71 σε ένα Μου λένε πως τελικά μπορούμε να ψήσουμε την 69 ως προσθήκη του κυρίου Ζασάδα. Υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. Τώρα στην 71. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να επαληθεύσουμε την 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Α, δουλεύει τώρα. Ωραία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 72 τεκάο υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Και ξεκολουθεί να δουλεύει το μηχάνημά σας. Ωραία. Πέρας. Απορρίπτεται. Εβδομήντα τρία υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική. F υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Εβδομήντα έξι σε ένα Πάλι είναι μια προσθήκη που μπορεί να ψηφιστεί χωριστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική G με ψηφοφορία σε δύο, σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο μέχρι το free of charge και μέρος δεύτερο μέχρι το booking. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτό, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές επίσης δεκτό. 91 και 92 Φώστερ Φαντάλεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Ήμκο 17 υπέρ. Κατά αποχές να την επαληθεύσουμε. Αρχιετή η ψηφοφορία. Δύο υπέρ. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. 99. Φόρτμαν κολ υπέρ. καταπίπτει εξαιτία της ΙΜΚΟ, της αντίστοιχη που ψηφίσαμε. 100 για την 10α, παράγραφο 10α, υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 12 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 101 Μαρτσίνκοβιτς υπέρ κατά. Ε, ποιοι, θέλουν να ψηφίσουν από τους σοσιαλιστές Μαρσίνκοβιτς υπέρ. Μπείτε στον κόπο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός H. Υπάρχει μία προφορική από τον κύριο Σασάντα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν όχι ψηφίζουμε απευθείας. Και υπάρχει και μία τμήματική που ζήτησαν οι πράσινοι σε τρία τμήματα, δηλαδή προφορική και τμήματική, για την υποτιθέμενη συμβιβασμό. Safely η πρώτη, μετά PRMs, μέχρι PRMs και η τρίτη τελειώνει στο modes. Λοιπόν, πρώτα η προφορική ζασάντα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα τα τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε το τρίτο. Εντάξει. Αρχίζει η ψηφοφορία για το τρίτο. Κράμερ υπέρ, δύο επιπλέον υπέρ που δεν έχουν κάρτα, πέρας 22, άρα εγκρίνεται. 107 προσθήκη υπέρ. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε. Την 107 αρχίζει η ψηφοφορία. Κράμερ και ο κύριος Κράμερ, δύο επιπλέον υπέρ, πέρας. Εγκρίνεται 25-22. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27. Ήμκο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός ΆΙ Ιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 121 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. 121 έλεγχος, αρχίζει η ψηφοφορία και δύο ψήφοι επιπροσθέτως. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, νομίζω ότι εγκρίνεται. Ελέγχουμε. Δύο επιπλέον υπέρ. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Ήμκο 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ήμκο 11. Ελέγχουμε και δύο κατά επιπροσθέτως. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβασμός J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 τσικάου με την προσθήκη που βλέπετε. In due time αντί good time υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 κόχ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός κάπα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε 141 ελέγχουμε αρχίζει η ψηφοφορία έχουμε και έναν υπέρ έναν κατά πέρας απορρίπτεται 143 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός L υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός M υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία για την 152. Έχουμε δύο επιπροσθέτως, υπέρ δηλαδή. Πέρας 24-21 εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία 153, ψηφίζατε όλοι. Έχουμε και μία αποχή και μία ψηφοκάτα. Πέρας εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 Φώστερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 158 βαντάλεν υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά αποχές μπορούμε να ελέγξουμε. 159 αρχίζει ο έλεγχος και έχουμε και δύο ψήφους κατά. Ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 14 υπέρ κατά Ελέγχουμε. ΙΜΚΟ 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Και έχουμε και δύο επιπροσθέτως υπέρ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την 160. Αρχίζει η ψηφοφορία με δύο ψήφους υπέρ, επιπροσθέτως, πέρας. Απορρίπτεται. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 164. Φώστερ. Α, όχι, καταπίπτει. Ήμκο 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169. Κόχ υπέρ. Κατά. Αποχές ε, ελέγχουμε παρακαλώ. 169. Αρχίζει η ψηφοφορία. και δύο, ένας μάλλον υπέρ, ένας κατά. Πέρας, εγκρίνεται. 170 συντακτικό καθαρά, ε, 20, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 173 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε όμως 177 αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είχαμε και έναν υπέρ, έναν κατά. Απορρίπτεται. 175 τσικάου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 καθαρά συντακτική τροπολογία. Κόσα, άρα δεν ψηφίζουμε. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 180. Αρχίζει η ψηφοφορία με δύο ψήφους υπέρ. Πέρας με δύο ψήφους ε, επιπροσθέτως χωρίς κάρτα. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε και πάλι 181. Νομίζω ότι είναι ίδιο το αποτέλεσμα, αλλά ελέγχουμε με δύο ψήφους υπέρ επιπροσθέτως. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 183 φιντάντσα υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 184 υπέρ, κατά, αποχές ε, έλεγχος παρακαλώ, ο οποίος και αρχίζει, 184 ένας υπέρ, ένας κατά, επιπροσθέτως, πέρας και απορρίπτεται. 182 κόσα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 24 κατά πίπτη παράγραφος 28 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να ελέγξουμε. Για την 3 αρχίζει η ψηφοφορία και έχουμε δύο ψήφους κατά χωρίς κάρτα. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε παρακαλώ. Τέιλο υπέρ. Ε, αρχίζει η ψηφοφορία, με συγχωρείτε, με δύο ψήφους υπέρ, χωρίς κάρτα. Πέρας. Εγκρίνεται. Πέντε Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έξι ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7, 8, 9, 10 παρόμοιες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά ελέγχουμε 14 αρχίζει η ψηφοφορία για την 14 και έχουμε 2 υπέρ χωρίς κάρτα. Πέρας εγκρίνεται 24 ψήφοι έναντι 22, 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται δύο Κόσα. Με την προφορική του εισηγητή όλοι είναι ευτυχείς με την προφορική υπέρ λοιπόν κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία η οποία και αρχίζει και έχουμε δύο υπέρ χωρίς κάρτα Κράμερ Ελκαντράουι πέρας 41 υπέρ και ένας μόνο κατά. Να συγχαρούμε τον κύριο Τέιλορ, εγκρίνεται η έκθεσή του. We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 από την Διεύθυνση Κλιματικών Αλλαγών. Νομίζω ότι έχει έρθει. Okay. Ah, yeah, thank you. Okay. Μάλιστα. Yeah, I'm going to go straight in anyway. <laughs> Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μαζί μας τον κύριο Τζος Ντέλμπεκε, Γενικό Διευθυντή για την δράση για το κλίμα, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Στη συνέχεια θα έχετε και εσείς δυνατότητα να πάρετε το λόγο. Κύριε Ντέλμπεκε, σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς επειδή ήρθατε εδώ. Ήρθατε και νωρίτερα, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε και νωρίτερα την παρουσίαση αυτή. Αν υπάρχουν ε, ορισμένοι που θα ήθελαν να αποχωρήσουν, ε, τότε ας το κάνουν για να ξεκινήσουμε. Κύριε Ντελιπέκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Είναι πραγματική ευχαρίστηση να βρίσκομαι εδώ. Θα σας ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την αεροπορία, τι κάνουμε με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και πώς εξελίσσεται διεθνώς όλη συζήτηση. Ξέρετε ότι οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν ένα πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που μας δίνουν πάρα πολλά επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια μεγάλη δέσμη κανονισμών για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, για τα αυτοκίνητα, για τις μονάδες παραγωγής ενέργειας. Ένας από τους τομείς όμως ο οποίος δεν καλύπτετο ήταν η αεροπορία και οι διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές. Ξεκινώντας λοιπόν με την αεροπορία, υπήρχε γενικότερη εντύπωση ότι θα έπρεπε και ο τομέας αυτός να καλυφθεί γιατί αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΚΑΟ μπορούμε να δούμε ένα 700% αύξηση τα επόμενα χρόνια και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι ενώ μειώνουμε τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα σε άλλου τομεί, αυξάνονται οι εκπομπέ αυτέ για τι αεροπορικέ μεταφορέ. Η αεροπορία αποτελεί βέβαια έναν διεθνή κλάδο, επομένω πρέπει να ληφθούν μέτρα πολιτική με τρόπο εντελώ διαφορετικό από ό,τι κάνουμε για παράδειγμα για τα οχήματα στην Ευρώπη ή για τι μονάδε παραγωγή ενέργεια. Τρει παρατηρήσει θα ήθελα να κάνω. Καταρχά, μια ιστορική αναφορά η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ανέκαθεν έλεγε ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, δηλαδή στον ΙΚΑΟ. Ο ΙΚΑ όμω δεν παρήγαγε πάρα πολλά αποτελέσματα, επομένω οι νομοθέτε και προφανώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άρχισαν να ανησυχούν ιδιαίτερα και ασκούσαν πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υποβάλει μια δράση ακόμα και σε περιφερειακό επίπεδο, εφόσον δεν υπήρχε κάποιο διεθνέ πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν το 2008 μέσω τη συναπόφαση εγκρίναμε έναν κανονισμό προκειμένου να συμπεριληφθεί η διεθνή αεροπορία στο σύστημα εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτή ήταν και η γραμμή που πήραμε και από τον ΙΚΑΟ, γιατί υπάρχουν δύο βασικές αρχές στον ΙΚΑΟ. Θεωρεί δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν φόροι ή εισφορές όσον αφορά την αεροπορία, αλλά ήδη από τις αρχές του 2000 ο ΙΚΑΟ είχε πει ότι ένα σύστημα σαν το δικό μας, το ETS, δεν αποτελεί ούτε φόρο ούτε εισφορά, είναι κάτι το διαφορετικό. Επομένως, Μερικές φορές συγχαίουμε το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών με ένα σύστημα φορολόγησης αλλά μπορούσε να γίνει αποδεκτό το ETS από τον ΙΚΑΟ. Επίσης, ο ΙΚΑΟ μας είπε ότι το μέσο αυτό ήταν ε, χρήσιμο, το να τεθεί δηλαδή ένα ανώτατο όριο στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο ΙΚΑΟ όμως δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ένα δικό του σύστημα, απλώς ενθαρρύνει τις περιφέρειες ή τα κράτη να ενσωματώσουν στα εθνικά του συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων την αεροπορία. Η απόφαση αυτή αεροπορια η αποφαση αυτη ληθηκε το 2004 και αυτό ακριβώ κάναμε και στην Ευρώπη. Επομένω, εγκρίθηκε μια νομοθεσία μέσω τη συναπόφασης το 2008 μέσω ομοφωνίας στο Συμβούλιο και με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα σε σημερινή κατάσταση όπου έχουμε σχεδόν εντελώς εφαρμόσει την νομοθεσία μας από την 1η Ιανουαρίου του 2012 αρχίζει να ισχύει η νομοθεσία αυτή. Από την ημερομηνία λοιπόν αυτή όλες ε, οι εκπομπές θα πρέπει να καλύπτονται μέσω του συστήματος δικαιωμάτων εκπομπών και αυτά τα δικαιώματα στη συνέχεια δίνονται δωρεάν, παρέχονται δωρεάν σε ένα πολύ μεγάλο, σε ένα πολύ ευρύ επίπεδο γιατί ξέρετε ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και σε περιφερειακό επίπεδο και ένα 85% των εκπομπών του 2012 θα καλυφθούν μέσω των ε, δικαιωμάτων εκπομπών δωρεάν και αυτό θα ισχύει για κάθε χρόνο από το 2013 και μετά. Επομένως, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να καλύψουν το εναπομείναν ποσοστό. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν βρισκόμαστε σήμερα. Ακολουθήσαμε την νομοθεσία όπως αυτή δημιουργήθηκε μέσω της συναπόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, ποια είναι η δική μας η θέση σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι η νομοθεσία αυτή αντιμετώπισε κάποια διεθνή αντίσταση και σε πολλές διμερείς επαφές πρέπει να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό και σε πολλές συνόδους επίσης. Και νομίζω ότι ένα σημείο καμπής ήταν η Σύνοδος Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένε Πολιτείε τον Νοέμβριο 2011 όπου εφήγει το ζήτημα αυτό και όπου τελικά είχαμε την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να ανοίξουμε και να συνεχίσουμε τις συζητήσεις στα πλαίσια του ΙΚΑ, του Διεθνού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορία. Έκτοτε, ο κύριος Κόμπε, ο, ο πρόεδρος του ΙΚΑΟ και ο κύριος Μπενζαμά, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΚΑΟ, έχουν αρχίσει να μιλάνε για την επιτάχυνση του προγράμματος εργασία του ΙΚΑΟ όσον αφορά τις ε, εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών. Επομένως, εμείς ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ θετικά σε αυτό, γιατί ανέκαθεν θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πολυμερής λύση και όχι μια περιφερειακή λύση στο πρόβλημα. Και ακολουθούμε ουσιαστικά τρεις βασικούς άξονες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν οποιοδήποτε σύστημα του ΙΚΑΟ αρκεί να μειώνει τις εκπομπές περισσότερο από ό,τι τα περιθωριακά ευρωπαϊκά συστήματα. Νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι ιδιαίτερα δελεαστικό, γιατί αναφερόμαστε σε ένα κλάδο που έχει διεθνή δραστηριότητα, επομένω ένα τέτοιο παγκόσμιο σύστημα θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει εκπομπέ των αεροπορικών μεταφορών. Μια άλλη βασική αρχή είναι το σύστημα αυτό να μην εισάγει διακριτικές μεταχειρήσει, διακριτική μεταχείριση με συγχωρείτε, ανάμεσα σε αεροπορικέ εταιρείε. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για τη δική μα ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα πρέπει να αποτελεί βασική αρχή για οποιοδήποτε σύστημα εγκρίνει ο ΙΚΑΟ. Δεν πρέπει να έχουμε διακριτική μεταχείριση ανάμεσα σε αεροπορικέ εταιρείε γιατί ξέρετε ότι στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για τις κλιματικές αλλαγές μιλάμε για τις κοινέ και διαφοροποιημένες ευθύνες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι βιομηχανοποιημένες χώρες θα πρέπει να κάνουν περισσότερες προσπάθειες. Εμείς δεν θέλουμε να εισάγουμε την ερμηνεία που έχει δοθεί από ορισμένου στις διαφοροποιημένες αυτές ευθύνες σε σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές. Ορισμένοι λέγανε ότι οι βιομηχανικές χώρες, οι, ε, χώρες θα πρέπει να κάνουν τα πάντα, ενώ οι, οι υπόλοιπε χώρες δεν θα πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη προσπάθεια. Θεωρούμε ότι αυτό στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και τάσεται κατά των αεροπορικών μεταφορών των διαφόρων αεροπορικών εταιριών. Η δεύτερη λοιπόν αυτή αρχή ήταν η αρχή των μη, της μη μεταχείρισης και τρίτον είπαμε ότι σε περίπτωση που ο ΙΚΑΟ καταλήξει σε ένα πλαίσιο δράσης και όχι ένα δικό του πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένα, συγκεκριμένοι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από πραγματικά μέτρα, διαφορετικά θα καταλήξουμε απλώς σε κάποιες καλές δηλώσεις, σε κάποιες θετικές προθέσεις, χωρίς όμως να πετυχαίνουμε ποτέ τους ε, στόχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στόχους, αλλά οι στόχοι αυτοί να συνοδεύονται και από συγκεκριμένα μέτρα. Αυτό καλύπτει λοιπόν το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω, ότι είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι στα πλαίσια του ΙΚΑΟ, ότι υπάρχει ήδη ένα πρόγραμμα εργασίας για τη συνεργασία με τον ΙΚΑΟ και συμβάλλουμε κι εμείς ε, πολύ ενεργά σε όλες αυτές τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες που θα πρέπει να διευθετηθούν και που θα βοηθούσαν τις δραστηριότητες του ΙΚΑΟ. Έρχομαι λοιπόν στο τρίτο σημείο τώρα. Στη Μόσχα είχαμε μια συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα, μια συνέχεια συνεδρίασης που έλαβε χώρα τον Νοέμβριο στο Δελχή και θα γίνει και στη Σαουδική Αραβία μια ακόμα επόμενη συνεδρίαση. Στη Μόσχα λοιπόν εγκρίθηκε μια δήλωση η οποία Μάλιστα ανακοινώθηκε και στο Διεθνή Τύπο. ενδεχομένω θα θέλατε να δείτε πώς ερμηνεύουμε εμείς ε, την δήλωση αυτή της Συνόδου της Μόσχας. Είμαστε κάπως απογοητευμένοι βέβαια, γιατί η δήλωση αυτή της Μόσχας είναι αυτό που θα ονόμαζε κανείς μια συμμαχία των μη πρόθυμων τελικά. Εμείς ε, ήδη πριν την ε, διοργάνωση της Συνόδου στην Μόσχα είχαμε πει ότι θα θέλαμε να καταλήξουμε σε μια θετική συμβολή, πώς θα καταφέρουμε δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι είμαστε κάπως απογοητευμένοι με, το, με την έκβαση της συνόδου αυτής, με την δήλωση που γίνεται προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές του θερμοκηπίου. Δεν ήταν τόσο θετική η δήλωση της ε, συνόδου της Μόσχας. Τι λέγεται όμως τη δήλωση αυτή παρουσιάζονται κάποιες εναλλακτικές λύσεις στη δήλωση αυτή. Εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει με την νομοθεσία της. Ορισμένοι θα μπορούσαν να πούνε ότι πρόκειται για μια δράση αστικά η οποία στρέφεται κατά της δικής μας της νομοθεσίας καθότι προτείνονται διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις ακόμα και για τον ΙΚΑΟ ο οποίος ήταν σε θέση να προτείνει κάτι διαφορετικό από αυτό που γίνεται τώρα. Το θετικό είναι ότι η δήλωση της Μόσχας, παρά τις συναλλακτικές αυτές λύσεις που προτείνονται, παρόλα αυτά λέει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την εργασία που γίνεται στα πλαίσια του ΙΚΑΟ. Και αυτά είναι, αν θέλετε, τα βασικά θετικά νέα τα οποία έχουμε στην συνάντηση της Μόσχας. Από ό,τι φαίνεται όλοι οι ενδιαφερόμενοι είναι σε θέση πλέον να εργαστούν στα πλαίσια του ΙΚΑΟ και νομίζω ότι αυτή είναι μια καταπληκτική ευκαιρία την οποία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Η δήλωση της Μόσχας υπογράφηκε από 23 κράτη. Δεν είναι ακριβώς τα κράτη αυτά τα οποία υπέγραψαν για τη δήλωση στο Δελχή. Ορισμένα κράτη ουσιαστικά δεν συμμετείχαν αυτή τη φορά στην ε, δήλωση αυτή και έχουμε και κάποια μικρά κράτη τα οποία μπήκαν στη λέσχη αυτή. Πέντε από τις 23 χώρες δεν καλύπτονται και από την νομοθεσία μας, γιατί η νομοθεσία μας δεν προβλέπει εφαρμογή σε αυτά τα κράτη. Το συμπέρασμα ουσιαστικά είναι ότι ότι οποιοδήποτε μέτρο τελικά και να υιοθετηθεί, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόλις αυτό εμφανιστεί η διακριτική μεταχείριση η οποία θα μπορούσε να εισαχθεί κατά των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή και εφόσον γίνει κάτι τέτοιο εμείς θα αναλάβουμε δράση αμέσως. Επίσης στην δήλωση της Μόσχας υπόθηκε κάτι κάπως διαφορετικά σε σχέση με τη σύνοδο στο Δελχή. Αναστολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας το ενδεχόμενο αναστολή αυτή διατυπώνεται με έναν τρόπο λιγότερο επιθετικό από ό,τι έχουμε στη δήλωση του Δελχή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την σύνοδο της Μόσχα. Το θετικό είναι ότι μπορούμε να έχουμε μια συνεργασία διεθνή όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Και το πιο θετικό βέβαια είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στα πλαίσια του ΙΚΑΟ, Επομένω, τι γίνεται τώρα στα πλαίσια του Διεθνού Οργανισμού Πολιτική Αεροπορία. Στι αρχέ ε, Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθο, 12 με 12 Μαρτίου, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο του ΙΚΑΟ και θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Η συνάντηση λοιπόν αυτή θα είναι σημαντική. Στη συνέχεια ελπίζουμε ότι ε, ο ικαό, όπως είχε υποθεί και στο παρελθόν, θα προτείνει ένα περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών λύσεων για τον περιορισμό των εκπομπών των διεθνών αεροπορικών μεταφορών μέχρι τον Ιούνιο και ότι θα επεξεργαστούν μέχρι το τέλος του έτους μία μοναδική εναλλακτική λύση θα πρέπει να τηρήσει ο ΙΚΑ το χρονοδιάγραμμα, αυτό, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, γιατί η δική μας προθεσμία, για τη δική μας την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ο Απρίλιο του 2013. Τον Απρίλιο του 2013 θα έχουμε την πρώτη ημερομηνία παραχώρησης, δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να παραχωρήσουν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια του ETS. Απρίλιο του 2013 λοιπόν η δική μας καταλεκτική προθεσμία, επομένω έχουμε μπροστά μας πάνω κάτω ένα έτος. Ένα έτος όμως για την δημιουργία νομοθεσίας είναι περιορισμένο χρονικό διάστημα. Χαιρόμαστε πάντως που βλέπουμε ότι επιταχύνει πλέον τις εργασίες του ο ΙΚΑΟ και τα πρώτα μηνύματα, τα πρώτα δείγματα, ουσιαστικά τις πρώτες ενδείξεις θα τις έχουμε στο Συμβούλιο του ΙΚΑΟ τον Μάρτιο. Εμείς λοιπόν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σαφώς υπέρ μιας διεθνούς παγκόσμιας λύσης για την μείωση των εκπομπών του νερίου θερμοκηπίου για την διεθνή αεροναυτιλία. Έχουμε το δικό μας περιφερειακό σύστημα, το ETS. Δεν πρόκειται να στείλουμε τη λειτουργία του συστήματος αυτού, πάντως είμαστε σε θέση να το τροποποιήσουμε εφόσον και αν ο ΙΚΑΟ προτείνει μια πραγματική παγκόσμια λύση, ένα πραγματικό διεθνές παγκόσμιο πρόγραμμα. Και η καταληκτική ημερομηνία που έχουμε θέσει είναι ο Απρίλιος του 2013. Ελπίζουμε πάντως ότι με την επιτάχυνση της εργασίας που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, ότι θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά διεθνές παγκόσμιο σύστημα μέσω του ΙΚΑΟ σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ήδη στην Επιτροπή μας είχαμε ζητήσει από την Κομισιόν να δει αυτό το θέμα εγκαίρως, να μην ευνηδιαστούμε όπως και με άλλα θέματα. Και ακόμη χειρότερο, και επανέρχομαι στην τελευταία παρατήρηση, ξαφνικά να λάβει μια απόφαση η Κομισιόν πριν πάει στην ε, συναπόφαση και να αποφασίζει μόνο με το Συμβούλιο και να μείνει απ' έξω το Κοινοβούλιο είχα μια τέτοια εμπειρία, δεν θα το αποδεχτούμε δεύτερη φορά, ειδικά σε αυτόν τον τομέα. Διεθνώ τώρα. Εάν μιλάμε για αεροπορία ή ναυσιπλοεία, είναι δύσκολο το θέμα. Εμείς παραμένουμε πεπισμένοι πως τα μέτρα τα οποία θέλουμε να περάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει ε, εκ των προτέρων να προσπαθούμε να έχουμε ε, διεθνή στήριξη για αυτά αντί να αναζητούμε εκ των υστέρων. Αυτό έχει δείξει εμπειρία. Και τελευταία παρατήρηση, ε, ερώτηση. Εάν, και όπως φαίνεται, δεν γίνει σε διεθνές επίπεδο αυτό το οποίο θέμε. Εάν στο επίπεδο του ΙΚΑΟ δεν υπάρξει πρόοδος, ποια μέτρα θα λάβει η Κομισιόν από το 2013 για τις χώρες και τις εταιρείες που δεν εκπληρώνουν αυτές τις απαιτήσει. Ε, ποια είναι τα δικά μας μέτρα, δηλαδή απέναντί τους, αντί να ρωτάμε ποια είναι τα αντίπεινα που λαμβάνουν οι άλλοι εναντίον μας. Ε, πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, μας απειλούν με ε, περιορισμούς στις υπερπτήσεις και τα λοιπά. Η Κομισιόν πώς τις βλέπει αυτές τις απειλές εντάξει, ότι θα κάνουμε κάτι και ότι είμαστε κατά είναι λογικό, αλλά με τις οικονομικές ζημίες που ήδη υπάρχουν, ε, τι θα γίνει. Και αναφέρουμε βέβαια σε τι προληπτικά μέτρα θα λάβετε. Ευχαριστώ κύριο Σαλχαντραουή για τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντελμπέκε. Βεβαίω, ε, πέρσι ακούγαμε διάφορες ε, ιστορίες ε, περίεργες για την οικονομικό αντίκτυπο από συναδέλφους από το Κογκρέσο που δεν ήταν καλά ενημερωμένοι για τον αντίκτυπο των μέτρων μας. Αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ πως θα πρέπει να πάμε σε δύο φάσεις. Πρώτα απ' όλα να προσαρμόσουμε νομοθεσία για τα ενδοευρωπαϊκά δρομολόγια για να τα συνηθίσει ο κόσμος ε, στο πώς ε, θα διαμορφωθεί η κατάσταση και μετά σε μια επόμενη φάση ε, να κατήψουμε όλο τον κόσμο. Αλλά πρέπει βεβαίως όσον αφορά και τη συναπόφαση να είμαστε και συνεπείς με τον εαυτό μας. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω κάποια ερωτήματα. Πρώτον, αναφερθήκατε στο τι γίνεται εντό του ΙΚΑΟ, που είναι πράγματι ουσιαστικό. Και θα πρέπει μετά να δούμε πώς θα αλλάξουμε την ομοθεσία μας. Πότε θα ολοκληρωθεί λοιπόν αυτή η διαδικασία, πότε θα μπορέσουμε να πούμε πως ναι εντάξει είμαστε έτοιμοι να είμαστε κάπως πιο ευέλικτοι και εάν πρέπει να γίνουν αυτές οι προσαρμογές, να ακολουθεί ολόκληρη διαδικασία της ε, συναπόφασης. Ε, αυτή χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρωθεί και από νομική σκοπιά ε, τον Απρίλιο του 2012 εάν έχει μια πρόταση ολοκληρωμένη ο ΕΚΑ φέτος. Επίσης αναφέρθηκε η δυνατότητα μία χώρα να λάβει συγκρίσιμα μέτρα. Έχετε ενδείξεις πως κάποιες χώρες πάνε προς αυτή την κατεύθυνση ή θα συζητηθούν τα πράγματα μόνο στο πλαίσιο του ΙΚΑΟ. Και σε αυτό το οποίο ε, είπε ο συνάδελφος, τι θα συμβεί σε περίπτωση που δεν έχουμε λύση, δεν θα αντιδράσουν όλες οι χώρες με τον ίδιο τρόπο. Οι άλλες θα λένε πως ε, θα λάβουμε αντίπεινα ή δεν πληρώνουμε. Τι θα γίνει με τα μέτρα λοιπόν που θα πρέπει να λάβουμε σε ευρωπαϊκό παιδί. γιατί αλλιώς θα καταλήξουμε σε μία κατάσταση αθέμητο ανταγωνισμό. Άλλες εταιρείε θα πληρώνουν και άλλε όχι. Και τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε για τη συνάντηση στη Ρωσία, πως δεν ήταν όλε οι χώρες, κάποιες χώρες, αλλά ήταν οι μεγάλες χώρες με αεροπορία, Ήπα, Ρωσία, Κίνα κτλ. Οπότε σημαντική, σημαντικό ποσοστό της αγοράς που δεν πρέπει να υποτιμάμε. Ε, δεν πρέπει να υποτιμάμε την, ε, την ε, αντίσταση δηλαδή. Πρόκειται, θεωρείτε εσείς ότι πρόκειται για, για μπλόφα ή για κάτι σοβαρό. Γιατί εσείς που παρακολουθείτε τα πράγματα λέτε πως οι χώρες αυτές που είναι κατά ε, μήπως αναζητούν μια λύση. Κυρία Μάισνερ, ναι ευχαριστώ. Πράγματι το εμπόριο των εκπομπών έχει λογική μόνο εάν ισχύει για όλα τα μέσα μεταφοράς και παγκοσμίω. Νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Το πρόβλημα είναι πώς θα το επιβάλλει κανείς κάτι τέτοιο. Και βλέπω πως είναι ενισχυτικά αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μόσχα. Εμείς υποτιμήσαμε ως Ευρωπαίοι τον ε, συνασπισμό των απροθύμων, όπως το είπατε. Αποφασίστηκαν ήδη νομίζω αντίπεινα για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Ε, ε, μιλάνε για απαγόρευση στην Κίνα. Και αν η και η Κίνα και η Ρωσία και η Ινδία όλες μαζί έχουν κοινή στάση, ε, είναι σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό για μένα θα μπο... τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, να ασκήσουμε επιρροή στον ΙΚΑΟ. Και νομίζω είναι καλύτερο, αντί να ερεθίζουμε τους άλλους ε, με τέτοιες ε, κινήσεις, να δούμε πώς μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε στον ΙΚΑΟ. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος, κατά την άποψή μου. Να σκεφτούμε το τι είπε ο Σαΐντ Χαντραουί. Πώς γίνεται βεβαίως από τεχνική σκοπιά με την ομοθεσία και πώς μπορούμε να πείσουμε και τους υπόλοιπους πως ε, η δική μας άποψη είναι σωστή. Γιατί εγώ ανησυχώ με αυτά τα οποία συνέβησαν στη Μόσχα και φοβόμουν ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά και να μην απομονωνόμαστε. Να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε και τις άλλες χώρες. Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ. Εγώ διαφωνώ. Εάν δηλαδή λέμε πως η Ευρώπη υποκύπτει στην πρώτη δυσκολία, έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας. Θα αφήσουμε όλα τα μέτρα τότε του κλίματος, είτε είναι κατά της βιομηχανίας, είτε είναι κατά των άλλων μέσων ε, ε, μεταφοράς. Εάν λέτε κυρία Μάισνερ πως πρέπει να είναι τα πράγματα όλα ίδια στα μέσα μεταφοράς, πρέπει τότε αμέσως και συνεπώς να σταματήσουμε ε, τα πάντα και στη βιομηχανία. Ε, μπορούμε να ξεχάσουμε την προστασία του κλίματος. Για τον ΙΚΑΟ δεν έχω καμία αισιοδοξία. Τι γίνεται τώρα εκεί μέσα. Οι ΙΠΑ έχουν κάνει συμμαχίες, μιλάμε για εκβιασμούς και αν λέμε άμα, μα, μα, μα, Παναγία μου», και θα σταματήσουμε να προστατεύουμε το κλίμα γιατί οι υπόλοιποι ε, το θεωρούν επιθετικό, ε, με συγχωρείτε. Πρόκειται πρώτον για ευρύτατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ξαφνικά ακυρώνεται και δεύτερον θεωρώ πως αυτό είναι αντίθετο με ε, πράγματα που έχουν αποφασιστεί, συζητηθεί σε άλλες παγκόσμιες ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό το οποίο εγώ θα έλεγα το οποίο δεν βλέπω, είναι πρώτον, ποιες είναι πραγματικά οι πιθανότητες να υπάρχει κάτι ανάλογο αποτελέσματος στον ΙΚΑΟ. Πέρα από τις ωραίες δηλώσεις ότι ίσως σε 100 χρόνια μπορεί να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Και πώς θα κρίνουμε το εάν ένα μέτρο είναι επαρκές. Δεν έχουμε συγκρίσιμα δίκτυα μέτρησης Εκεί πέρα έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Τι γίνεται με την αμοιβαία ε, αναγνώριση των αποτελεσμάτων μέτρηση, όσον αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, τι εκπομπέ. Ε, εδώ πέρα παγκοσμίω δεν υπάρχει κάτι το συγκρίσιμο. Και βεβαίω μα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όταν μιλάμε για αντίπεινα δηλαδή. Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα αντίπεινα. Τα αντίπεινα, κατά την άποψή μου, πρέπει να, να τα δούμε πρώτα απ' όλα, γιατί ε, εντάξει, είναι και λίγο θεατρινισμοί αυτά τα πράγματα. Έχουμε περιφερειακές αγορές και συνδέσεις μεταξύ τους Για αν μιλάμε για εκβιασμούς κατά της Ευρώπης μπορούμε να απαντήσουμε. Πώς υπολογίζεται λοιπόν αυτό σε σχέση το ένα με το άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ. Εμείς δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε ούτε τις αναπτυσσόμενες χώρες, ούτε τις είπα. Είναι σαφές. Αλλά αντιστρόφως και αυτοί δεν μπορούν να μας εξαναγκάσουν. Να πετάξουμε από το παράθυρο σας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μα απειλεί κάποιο. Γιατί ένα είναι σαφέ. Ακόμα και αν αυτό ο συνασπισμό των ε, απροθύμων ε, μειωθεί, κάποιοι θα παραμείνουν. Και βεβαίω ε, για τους σκεπτικιστές για το κλίμα στην Ευρώπη που λένε διάφορα θα μας λένε πως η υψή περιοχή του κόσμου είναι έξω οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. θα έχουμε αυτό το πρόβλημα γενικώ. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, το πρώτο βήμα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ποια αντίπεινα μπορούμε εμείς να λάβουμε εάν είναι να μιλήσουμε για αντίδραση της Ευρώπης. Τώρα να είμαστε προετοιμασμένοι. Όχι να λέμε «Ω Θεούλη μου θα πούν οι άλλοι όχι». Όχι μόνο για ζητήματα του κλίματος, για όλα τα ζητήματα σε οτιδήποτε ε, αφορά ε, τις εξωτερικές επιδράσεις των συγκοινωνιών. Το επόμενο σας το λέω, είναι στην αυτιλία και τα καύσιμα. Το μεθεπόμενο μετά στις ποτάμιες συγκοινωνίες κτλ. Εμείς, η Ευρώπη δηλαδή, γονατίζει αμέσως όταν, απαιτήσει κάτι, όταν απαιτήσουν κάτι οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά Αντιστρόφως όταν μιλάμε για το να προασπίσουμε τις δικές μας αξίες δεν συμβαίνει τίποτα. Και αμέσως πάρα πολύ εντός της Ευρώπης είναι πρόθυμοι να ακούσουν τις Ηνωμένε Πολιτείε όταν είναι κατερνητικό. Suspect... Κυρία Φώστερ, φαντάζομαι θα έχετε αντίθετη γνώμη. Ψυχανεμίζομαι. Ναι, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ε, αφήνω την κυρία Λίχτενμπερκ τα σχόλιά της και θα ασχοληθώ με τα δικά μου. Ε, ευχαριστούμε την Επιτροπή, μάλλον όχι την Επιτροπή, τον εκπρόσωπο για την ενημέρωση, αλλά για να είμαστε σοβαροί. Ε, νομίζω όμως ότι επικαιροποιήστε Θέλω να σας πω κύριε Ντελμπέκε ότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μας παράτησε εδώ και πολλά χρόνια ε, όταν προέβαλε το ETS. Δεν μιλώ για το ETS καθε αυτό, αλλά για το γεγονός ότι είχε προειδοποιηθεί η Επιτροπή από τη βιομηχανία, από διάφορους φορείς, ανθρώπους, πολιτικούς, από τα κράτη-μέλη, ότι θα ήταν κάτι το πολύ δύσκολο. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε φορολογία σε τρίτες χώρες. Μιλήστε για τέλη ή ό,τι θέλετε. Πρόκειται για μία φορολόγηση που δεν ήταν εφικτή. Γι' αυτό οι τρίτες χώρες δεν προσετερίστηκαν αυτή την ιδέα. Προχώρησαν με την μεγαλεπίβολη ιδέα τους και φτάσαμε σε αποκαίδια τώρα. Είπατε ότι το συζητήσαμε και τώρα προχωρούμε. Μιλάτε για αντίστοιχα μέτρα. Ποιος ε, αποφασίζει, εσείς είσαστε και δικαστής και κατήγορος και ένορκη. Όπως ξέρετε ότι 160 χώρες απέστειλαν μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγοντας εσείς κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά μη μας βάλετε σε αυτό το σχέδιο, εμείς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εσείς όμως είπατε στο Κοινοβούλιο, α όχι θαυμάσια, το ελέγξαμε, είναι νόμιμο, δεν με ενδιαφέρει τι λέει το ΔΕΚ, γι' αυτό είμαστε στο σημείο αρχής Μιλάμε για Βραζιλία, Ινδία, Κίνα, Αμερική, οι οποίοι υποτίθεται θα προσχωρήσουν, μα ξέρετε ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ ήμουν στην Ουάσιγκτον το καλοκαίρι, ξέρουμε τι κάνουν και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι δεν θα επιτρέψουν τους αερομεταφορείς τους να πάρουν μέρος σε αυτό το σχέδιο. Γι' αυτό μη μας κοροϊδεύετε. Το ξέρετε και εσείς και εγώ, διότι οι επιπτώσεις είναι πολύ ευρύτερες όταν μιλάμε για την βιομηχανία, για το εμπόριο. Δηλαδή πολλά ε, γελία, γελία ζητήματα θα είχαν αποφευχθεί. Είμαι κατηγορηματική. Είμαι στα όρια της αποπληξίας το γεγονός ότι μιλάτε για μια διαδικασία η οποία θα εισαχθεί. Τι θα γίνει εάν υπάρχουν ε, ε, πιστώσεις, εάν γίνεται πίστοση ε, για διοξίδιο του άνθρακα, για εκπομπές, πού πάνε τα χρήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να δοθούν. Άρα, μιλάτε για αντίπεινα από τρίτες χώρες. Μα εσείς το είχατε πει πρώτη, γιατί η κυρία Χέντεγκάρτ ήρθε σε αυτή την επιτροπή και μίλησε πρώτη για αντίτυπα. Δηλαδή, τι, πού θα φτάσουμε. Δηλαδή, αν οι Κινέζοι που είναι εντάξει, δεν προσχωρούμε, τι θα κάνετε. Βρισκόμαστε σε ακόμα χειρότερη θέση. Δεν ξέρουμε πού θα προχωρήσουμε και πώς. Γιατί να προχωρήσουν αυτές οι χώρες προς αυτό το σχήμα. Είτε εμεί το θεωρούμε σωστό είτε όχι. Γιατί. Γιατί να κινηθούν προς εμάς. Δεν μπορούμε εμείς να το παίζουμε ο δικαστή, Δηλαδή δεν δεχόμαστε, ε, δεν δέχονται οποιοδήποτε ε, τρόπο επιβολής σχεδίων, όπως δεν θα δεχόμασταν και εμείς από ε, Ρώσους, από Κινέζους. Θα λέγαμε και εμείς αντιστοίχως, εμείς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Δεν θα μας το επιβάλλουμε. Μιλάτε για ε, ε, θέμα αμοιβαιότητας και λέτε μετά «Α, δεν καταλαβαίνουμε γιατί οι τρίτες χώρες δεν προσχωρούν». Μα ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Άρα, όλα αυτά ξεκίνησαν τον Ιανουάριο, αλλά εγώ εκπροσωπώ τις επιχειρήσεις, ελπίζω μαζί με τον πρόεδρο, δηλαδή μας ενδιαφέρουν τα συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας και του, της Ευρώπης. Δεν μιλάμε μόνο για τους αερομεταφορείς. Μιλάμε για το, την αλυσίδα προμήθειας, μιλάμε για το διάστημα, μιλάμε για όλους τους φορείς. Άρα μιλάμε για θέματα ανταγωνισμού. Διότι θα υπάρχουν επιπρόσθετα τέλη και δαπάνες. Αλλά δεν υπάρχει συμφωνία από τις τρίτες χώρες, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Ε, η, η ΚΑΟ έχει 191 χώρες μην το ξεχνάτε αυτό. Θα συζητάμε και θα συζητάμε. Αλλά τώρα μιλάμε για ανταγωνισμό. Άρα θα υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και για τη βρετανική. Άρα η ρύθμιση δεν μπορεί να ισχύσει. Μιλάτε για μια ρύθμιση που θα ισχύει για όλους. Μα δεν θα ισχύσει για όλους γιατί οι τρίτες χώρες δεν θα προσχωρήσουν. Άρα μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό. Δηλαδή ποιο είναι το plan B τώρα θα ήθελα να μου πείτε. Η κυρία Διβεράκ. Ευχαριστώ. Περάσαμε την ε, μοιραία ημερομηνία της πρώτης πρώτους, του πρώτου του 2012. Όπως είπατε κύριε Γενικέ, οι επικρίσεις συνεχίζουν, συνεχίζονται παρά είστε αισιόδοξο σε σχέση με την εισήγησή σας και το μήνυμά μου είναι παρόμοιο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για την ε, εισδοχή του συστήματος των αερομεταφορέων στο σύστημα ETS, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη δήλωση του ΕΚΑΟ που μίλησε για μη δεσμευτικό πλαίσιο, μίλησε για διάλογο με τρίτες χώρες, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, μία συλλήβδην απόρριψη η θέση της Μόσχας την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί μιλήσατε για χώρες που έχουν κακή προαίρεση, η θέση λοιπόν αυτή δεν είναι αποδεκτή. Μιλήσαμε για εμπορικές εμπορική σύραξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως θέλουμε οι αερομεταφορείς να τηρούν το, τους κανονισμούς μας, όπως κάνουμε και εμείς τις υπερατλαντικές ε, πτήσεις. Ίσως η θέση μας ε, φαίνεται αμετακίνητη, αλλά αυτό αφορά και τους εταίρους. Και μπορούμε να μπούμε σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν θα οδηγήσει πουθενά. Ας καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και ας φτάσουμε σε λογικές θέσεις για όλους. Όπως είπε και ο Γενικός την προηγούμενη εβδομάδα, δεν θα πρέπει παρά να έχουμε μία πιο καθαρή αεροπλοεία και πιο διαφανή. Και δεν θα πρέπει να πλήξουμε την αεροναυσιπλοεία όπως έγινε τέσσερα χρόνια πριν. Θα, θα πρέπει να φτάσουμε σε μία ε, γενικά αποδεκτή θέση χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τους αερομεταφορείς μας. Ε, δέχομαι τις θέσεις της Επιτρόπου Χέντεγκάρντ την προηγούμενη εβδομάδα που κατήγγειλε τις τρίτες χώρες που αντιτάσσονται συλλήβδιν σε αυτό το σχέδιο αλλά που δεν προέβαλαν μία άλλη εναλλακτική θέση υπέρ του περιβάλλοντος. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τις θέσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ για να φτάσουμε στον κοινό μας στόχο. Κράμερ. Κυρία Φώστερ, δεν ξέρω αν είναι βρετανικό συμφέρον να υπάρξει ε, κλιματική αλλαγή και να βουλιάξει η μισή Μεγάλη Βρετανία. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η στρατηγική σας, συνεχίστε. Αλλά είναι άλλο το θέμα εδώ πέρα. Πρέπει να σταματήσει η κλιματική αλλαγή. Και έχουμε διαφορετικά προβλήματα. Και είναι, ε, κατά τα λοιπά, αδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναλόγως ε, αντιδρά. Ανεβάζουν τις τιμές για την υπέρπτυση της ε, Σιβηρίας οι Ρώσοι και εμείς απλά πληρώνουμε. Γιατί περνάνε οι Ρώσοι πάνω από την Ευρώπη ατιμόρυτα. Να ανεβάσουμε και εμείς τιμές. Βλάπτει τον ανταγωνισμό αλλά όχι προς το συμφέρον των ρωσικών εταιριών. Επίσης νομικά τα πράγματα είναι ε, ξεκάθαρα. Υπήρξε μια απόφαση για Αμερικάνοι τώρα Ρώσοι Κινέζοι δεν ασχολούνται με τα λεφτά. Μιλάμε για ψίχουλα. Το θέμα τους είναι ότι δεν θέλει να τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι να κάνουν. Αλλά εδώ πέρα ζουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι πελάτες αυτών των εταιριών. Αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό δεν πρέπει να εμφανίζεται ασθενή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυνατότητες. Γι' αυτό σας ρωτάω ξεκάθαρα ποιο είναι το σχέδιο Β εδώ πέρα. Και γνωρίζετε πως ε, το έχουν δεχτεί οι ευρωπαϊκές εταιρείε γιατί φοβόντουσαν πως θα καταργηθεί το αφορολόγητο των αεροπορικών καυσίμων που είναι πολλαπλάσιο το κόστος τότε. Αλλά δεν άκουσα από κανέναν επίτροπο να λέει αν δεν γίνει αυτό θα φορολογήσουμε τα καύσιμα. Η συμφωνία του Σικάγου λέει πως αυτή, το καύσιμο που είναι μέσα στο αεροπλάνο δεν μπορεί να φορολογηθεί. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν φόρο στα καύσιμα, αν πληρώναν και τα αεροπλάνα, τότε θα είχαμε αυτομάτως κανένα πρόβλημα. Όποιος ανεφοδιάζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα το πλήρωνε. Και να πει και η Κομισιόν, άμα δεν το θέλετε εντάξει θα κάνουμε και εμείς το άλλο. Θα λάβουμε μέτρα τα οποία θα προστατεύσουν το κλίμα, βεβαίως θα κοστίσουν λεφτά, πολύ περισσότερα θα εισπράξουμε έτσι και να μην υπάρχει και στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ αεροπλάνου και τρένου. Οπότε συγκεκριμένα το ερώτημά μου είναι ποια είναι η άποψη, το συζητάνε αυτό καθόλου ή είναι ταμπού παρά το ότι έχει το δικαίωμα η Ευρώπη προτιμάτε να μην το κάνετε. Κύριε Φαντάλεν, κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω λέγοντας πως στηρίζω το σύστημα εμπορίας των εκπομπών. Θεωρώ πως είναι ένα καλό σύστημα για να καταλήξουμε σε περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και βελτίωση της κατάστασης. Γιατί κάποιοι εδώ πέρα λένε πως έχει δημιουργήσει προβλήματα. Να σας υπενθυμίσω πως το 2008 έλαβε ομόφωνη απόφαση το Συμβούλιο και την ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία το Κοινοβούλιο. Οπότε τώρα τα δάκρυα που κυλάνε είναι κροκοδίλια. Πρώτον. Δεύτερον, για εμένα αυτό το οποίο βλέπουμε πλέον είναι η αποκάλυψη του Μπάρακ Ομπάμα. Πολλοί άνθρωποι τον θεωρούσαν σωτήρα, ηγέτη κτλ. κτλ. Αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι πως ο κύριος Ομπάμα όταν μιλάμε για πραγματική ουσία επιλέγει τα δικά του συμφέροντα και το περιβάλλον, για το περιβάλλον φτάνουν απλά τα ωραία λόγια. Και μιλήσατε πράγματι για την συμμαχία των προθήμων υπό την ηγεσία, υπό την ηγεσία του κυρίου Ομπάμα. Τώρα, θεωρώ πως ο Γενικός Διευθυντής είναι πράγματι ε, υπεραισιόδοξος. Επικρατεί ψυχρός πόλεμος αυτή τη στιγμή στον ε, ΙΚΑΟ. Ε, αυτό το οποίο υπάρχει μόνο είναι ωραίες δηλώσεις, αλλά ένα σύστημα το οποίο θα είναι τελείως ανεπαρκές. Οπότε το πρόβλημα ποιο είναι. Θα έχουμε εμπορικό ε, πόλεμο. Ο ΔΕ Γενικός Διευθυντής είπε πως ε, αμέσως θα λάβει η Κομισιόν αντίπεινα και διακριτικά μέτρα. Ε, αυτό είναι εμπορικός πόλεμος. Και βεβαίως αυτά τα είπε δημοσίως. Αλλά το ερώτημά μου εμένα προς τον κύριο Γενικό Διευθυντή είναι πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε έναν εμπορικό πόλεμο. Γιατί έχουμε να διαλέξουμε εντάξει, μεταξύ σκύλα και χάριβδης. Ναι, πρέπει να εισαχθεί το σύστημα, από την άλλη βεβαίω αν έχουμε ε, να μας απειλεί ένα εμπορικό ε, πόλεμος, δεν ξέρω, πρέπει να χαράξει μια ασφαλή πορεία μεταξύ των δύο οικομισιών. Κυρία Βόρτμαν Κόλ, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θυμάμαι καλά τις ε, συζητήσεις... Ε, μετά την ε, στήριξη που εκφράσαμε και ψηφίσαμε για το σύστημα εμπορίας εκπομπών για την αεροπορία. Και αναφέρομαι στην στήριξη που δώσαμε για μία οδηγία που συμπεριλαμβάνει τα ισοδύναμα μέτρη. Και ο Επίτροπος Ντάλι ήρθε εδώ πέρα όλος ελπίδες και μας δημιούργησε προσδοκίες πως η κατάσταση θα μπορούσε να επιληθεί. Πρέπει να το τονίσω αυτό το πράγμα. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα είχαμε σκεφτεί. Και από ό,τι φαίνεται στη Μόσχα οι άλλες χώρες προτίμησαν να μην συνεργαστούν αλλά να α, ε, αντισταθούν και τώρα άρα έχουμε μια απειλή για τον τι ευρωπαϊκέ αεροπορικέ εταιρείε. Μα δεν θέλαμε εμεί αυτό το πράγμα. Εμεί θέλαμε να αντιμετωπίσουμε το κλίμα, αλλά θέλαμε και ίσο ανταγωνισμό και αυτό εξακολουθεί να είναι η στάση της ε, Κομισιόν, ίση αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών ε, αεροπορικών εταιριών με τι άλλε εταιρείε του υπόλοιπου πλανήτη. Οπότε το θέμα τώρα θα είναι ποια θα είναι τα ισοδύναμα μέτρα. Γιατί ε, βλέπω δεν επιτυχάνουμε αυτό το οποίο θέλαμε να επιτύχουμε. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν πως είστε ε, έτοιμος πιθανώς να αλλάξετε την νομοθεσία ή την ερμηνεία της νομοθεσίας, αλλά ισοδυναμία δεν βλέπω. Ισοδυναμία πρέπει να έχει δύο πλευρές. Είτε οι άλλες χώρες θα, θα προσαρμοστούν στα δικά μας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά απίθανο, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, ή θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στον ΙΚΑΟ, αλλά αυτό σημαίνει πως πρέπει να υπάρξει ισοδυναμία για τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες. Να αλλάξει η δική μας ε, στάση. Είστε έτοιμος για κάτι τέτοιο. Γιατί κάποιοι συνάδελφοι εδώ πέρα μιλάνε εύκολα για ε, εμπορικούς πολέμους. Ένα καιρό οικονομικής κρίσης που δεν συμφέρει κανέναν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν η Κομισιόν ε, τι κάνει να προετοιμαστεί. Πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να προσαρμοστούμε. Γιατί ο καιρός, ε, ο χρόνος αρχίζει να πιέζει. Οι αεροπορικέ εταιρείε είναι εταιρείε και προετοιμάζονται ήδη για να αρχίσουν να πληρώνουν στο μέλλον και οι ανταγωνιστές τους όχι. Και σε καιρό οικονομικής κρίσης πραγματικά έχουμε μαύρα σύννεφα πάνω από τις αεροπορικές εταιρείε και τις θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ. Bradburn. Uh, thank you, Chairman. Well, I, I... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα λοιπόν τη συζήτηση αυτή και μου δημιουργείται εντύπωση ότι τα έχουμε ξαναδεί όλα αυτά. Θα ξέρετε κι εσείς κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε την πορεία της πρότασης αυτής, έχετε δει την όλη εξέλιξη και θυμάμαι στις συζητήσεις που κάναμε στο παρελθόν στην Επιτροπή μας, λέγαμε τότε ότι το σύστημα αυτό ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Για τους λόγους αυτούς ακριβώς που ακούσαμε και σήμερα. Είναι σαφές ότι όταν συζητήσαμε το σύστημα αυτό, ζούσαμε σε ένα διαφορετικό κόσμο, τουλάχιστον σε ένα διαφορετικό οικονομικό κόσμο. Ήταν πριν την οικονομική κρίση του 2008, πριν από την κατάσταση που έχουμε τώρα, όσον αφορά τα προβλήματα που έχουμε τουλάχιστον παγκοσμίω. Και άκουσα την όλη συζήτηση, είδα και άκουσα τα ίδια επιχειρήματα, ακριβώ τα ίδια επιχειρήματα τα οποία εκφράστηκαν και στην πρώτη συζήτηση που έγινε για την πρόταση αυτή. Ο κόσμο όμω έχει αλλάξει. Ο κόσμο έχει αλλάξει όχι μόνο εξαιτία οικονομική κρίση, αλλά και επειδή δεν νομίζω ότι την εποχή εκείνη ότι οι υπεύθυνοι καταλάβαιναν τις επιπτώσεις που θα έχει το σύστημα αυτό στην προσπάθεια να επιβάλλουμε το δικό μας σύστημα σε τρίτες χώρες. Σας είχα προτοποίησει τότε γι' αυτό. Η οικονομική πραγματικότητα κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οτιδήποτε και να πιστεύουμε για τις κλιματικές αλλαγές, η οικονομική πραγματικότητα τελικά αλλάζει τα πράγματα. Και όσον αφορά την οικονομική πραγματικότητα, εγώ βλέπω ότι υφίστανται οι ε, ίδιες ε, συνθήκες και περιστάσεις ε, όσον αφορά τον κλάδο αυτό όπως και σε άλλους. Το τμήμα αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όποτε προσπαθεί να κάνει κάτι προτείνει μέτρα τα οποία θα έχουν επιπτώσεις παγκοσμίω. Πρόσφατα είχαμε ανάλογες περιστάσεις την πρόταση εκείνη όσον αφορά την ποιότητα των καυσίμων που θα έχει αντίκτυπο στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν νομοθετεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλά, όταν προσπαθούμε όμω να επιβάλλουμε τη δική μα νομοθεσία στο εξωτερικό, τότε προφανώ θα αντιδράσουν και δικαιολογημένα κατά την άποψή μου. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα στο μέλλον. Πολλοί ομιλητέ είπαν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε στα πλαίσια του ΙΚΑΟ. Πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα, το δέχομαι. Αυτό είναι το κατάλληλο μέρος όπου θα πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε εμείς εδώ μονομερός να επιβάλλουμε σε άλλους. Και αν τελικά στα πλαίσια του ΙΚΑΟ καταλήξουμε σε μια λογική λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, τότε εγώ θα είμαι ο πρώτο ο οποίο θα χαιρετήσω την πρόοδο αυτή. Αλλά στην υφιστάμενη κατάσταση δεν νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς εδώ στην Ευρώπη, πώς θα αντιδράσουμε στην κατάσταση αυτή. Θα συνεχίσουμε σαν μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα εθελοτυφλούμε, θα φέρνουμε τελικά τις δικές μας αεροπορικές εταιρείες σε πολύ δεινή ανταγωνιστική σχέση σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες. Νομίζω ότι το πρώτο λογικό πράγμα το οποίο πρέπει να κάνουμε, κατά την άποψή μου κύριε Πρόεδρε, είναι να στείλουμε την Ευρωπαϊκή Αυτομοθεσία μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε κάποιες λογικές συμβαστικέ λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Κύριε Μπράτμπορν, συγγνώμη, σας αποκάλυψα Μπράντμπορη. Κύριε Μπράτμπορν, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Θα μιλήσω λοιπόν και εγώ και θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, γιατί στο παρελθόν με είχαν κατηγορήσει για διάφορα πράγματα και πολλές φορές όταν προσπαθεί κανείς να βοηθήσει μπορεί ακόμα και να τον καταγγείλουν, να τον κάνουν επίθεση. Επομένω εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία στα οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι. Η κυρία Ντεβεράκ αναφέρθηκε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο στον οποίο βρισκόμαστε. Έχει δίκιο. Άλλοι αναφέρθηκαν σε εμπορικό πόλεμο. Είναι και αυτό μία πιθανότητα. Αν δούμε επίση ε, και τα σενάρια που έχουμε μπροστά μας, μου κάνει πραγματικά εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο απορρίπτεται τις ε, χώρες αυτές ε, οι οποίες συμμετέχουν στην, στον περίφημο συνασπισμό των απρόθυμων. Ορισμένες, ε, ορισμένοι λένε ότι υπάρχουν κάποιε μεγάλε χώρε, οι ή κάποιες μικρές χώρες οι οποίε έχουν συμμετέχει. Έχουμε όμω τη Ρωσία, τι ΗΠΑ, την Ινδία, τη Σαουδική Αραβία και την Βραζιλία. Αυτέ είναι μεγάλε χώρε, τεράστιε χώρε. Όταν λοιπόν ε, συμφωνούν και συζητούν οι χώρες αυτές, τότε πρέπει να ακούσουμε τι έχουν να πούνε. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα αυτή τη στιγμή. όσον αφορά τις χώρες αυτές. Αν δείτε τι κάνουν συλλογικά και ουσιαστικά θα, δεν θα πρέπει να δικήσουμε την κυρία Χέντεγκάρτ γιατί για πρώτη φορά από τον τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουμε πλέον κάποιον που μπορεί να φέρει μαζί τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα να συμφωνήσουν οι τρεις αυτές χώρες για κάτι ενδεχομένως να πρέπει ε, να την στείλουμε και στη, στα Ηνωμένα Έθνη. Ενδεχομένως και εκεί να καταφέρει να κάνει κάτι για τη Συρία. Κατάφερε όμως να πετύχει το τεράστιο αυτό επίτευγμα. Να φέρει αυτούς τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές σε ένα κοινό τραπέζι συζήτησης και να συμφωνήσουν. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε και σαφώς το Κοινοβούλιο έχει τη δική του τη θέση. Θυμάστε τότε την έκθεση Γερζεμπόφσκι. Είχαμε πει τότε ότι μπορεί να υπήρχαν προβλήματα. Το βασικό όμω λάθο επιτροπή αυτή πριν από έξι χρόνια είναι ότι δεν ζητήσαμε τον κανόνα υπαριθμό 50 όπου επιτρέψαμε σε άλλες επιτροπές, όπως για παράδειγμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, χωρίς να υπάρχει ίδια μεταχείριση για όλες τις επιτροπές. Αυτό ήταν το μεγάλο θεμελιώδε λάθο που κάναμε τότε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, σε ένα σημείο καμπή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορεί να υποχωρήσει απλώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά αυτό το σχέδιο Β, η εναλλακτική λύση, δεν είπατε, κύριε Ντελμπέγκε, και ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε σε αυτό. Τι θα κάνετε, δεν είπατε τι θα κάνετε, πώς θα αντιδράσετε, αν τελικά τα κράτη αυτά λάβουν αντίμετρα, προχωρήσουν σε αντίπεινα. Και μην μου πείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει ουσιαστικά να μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό, γιατί αυτό, αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο Β. Φοβάμαι ότι προχωράμε σιγά σιγά σε μια κατάσταση όπου ενδεχομένως να βρεθούμε στο σημείο αυτό που τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν αποφασιστικά όσον αφορά την απόφαση αυτή. Η Κίνα, για παράδειγμα, μπορεί να πει ότι δεν θα πληρώσουν οι δικές μας αεροπορικές εταιρείε. Δεν θα περνάμε από τα αεροδρόμια σας. Και ενδεχομένως αυτό ακόμα και να επεκταθεί και στην αυτοβιομηχανία με τους κινητήρες Rolls για παράδειγμα. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να πω ότι στους ανθρώπους που εργάζονται σε ένα εργοστάσιο της Rolls Royce ότι κοιτάξτε, σώσαμε το εργοστάσιό σας αλλά δεν θα υπάρχει πλέον παραγωγή. Θα μπορούν να υπάρχουν διάφορες τοποθετήσεις, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια λογική θέση, να φύγουμε από τις ακραίες θέσεις. Μια λογική θέση για ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν θεωρώ ότι έχει αντιμετωπίσει ακόμα σωστά αυτή η Επιτροπή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και έχω και εγώ το δικαίωμα να εκφράζω αυτή την προσωπική άποψη, όπως και εσείς εκφράζετε τη δική σας την προσωπική άποψη. και δεν σα διακόπτω εγώ ποτέ, επομένω μην με διακόπτετε και εσεί, παρακαλώ πολύ. Ο κύριο Βαντάλε είπε επίση κάτι πολύ σωστό. Δεν νομίζω ότι η αλλαγή α, καθεστώτος στην Αμερική θα κάνει οποιαδήποτε αλλαγή, είτε έχουμε δημοκράτες είτε ρεπουμπλικανούς, το ίδιο, θα έχουμε την ίδια προσέγγιση και προφανώς στην Κίνα θα έχουμε αλλαγή καθεστώτο. Δεν νομίζω όμω ότι θα έχουμε αλλαγή όσον αφορά την προσέγγιση στον φάκελο αυτό. Αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή κατάσταση. Φτάνουμε κοντά σε έναν εμπορικό πόλεμο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φλούμε απλώς. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Ντελμπέκη. Μας είπανε πριν από πολλά χρόνια ότι θα έχουμε διαθέσιμους πόρους από το σύστημα αυτό που θα δοθούν στην έρευνα όσον αφορά τους κινητήρες της αεροναυτιλίας. Έτσι μας πουλήσετε το πρόγραμμα αυτό. Βέβαια, οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα έχουν πέσει πάρα πολύ, δεν μπορούμε τελικά να βγάλουμε χρήματα από το όλο σύστημα, επομένως τι θα κάνουμε στο μέλλον, πώς θα καταφέρουμε να ενθαρρύνουμε την έρευνα, θα μειώσουμε την ελεύθερη απονομή αυτών των δικαιωμάτων, πώς ακριβώς θα συλλέξουμε τους πόρους που θέλουμε και τι θα γίνει στη συνέχεια. Θα μπούμε και στον τομέα της βλέπετε για το μέλλον. Πρέπει να προχωρήσουμε σωστά με διεθνείς συμφωνίες. Διαφορετικά θα βρεθούμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα με τον IMO και με τις θαλάσσιες μεταφορές. τα ίδια ακριβώ προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε τι θαλάσσιε μεταφορέ όπω ακριβώ αντιμετωπίσουμε τώρα στα πλαίσια τη αεροπορία. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει μου. Σα είπα ότι είναι προσωπικέ μου απόψει. Πιστεύω όμω ακράδαντα ότι ε, βρισκόμαστε σε μια πολύ μπλεγμένη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και ολοκληρώνω με αυτό. Κύριε Ντελμπέκ, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τα ποικιλόμορφα σχόλια, για τα ποικίλα σχόλια και προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα. Νομίζω ότι πραγματικά έχουμε να κάνουμε με ένα ε, θέμα καθαρά ε, λογοδοσίας γιατί η κλιματική αλλαγή είναι ένα θέμα που αναγνωρίζουν όλοι και η Κίνα και η Ρωσία και όλοι οι παρόντες και νομίζω ότι οι διαπραγματεύσει των Αμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές αφορούν όλους τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και ε, ο ΙΚΑΟ επίσης έπρεπε και, ε, και εκείνος να συνεισφέρει. Έχουμε και έχουμε δύσκολες συζητήσεις για να μειώσουμε τις εκπομπές στον τομέα του αυτοκινήτου, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και της αεροπλοείας ε, γιατί ξέρουμε ότι οι εκπομπές θερμοκηπίου θα αυξηθούν επί 7 μέχρι το 2015. Αυτό λοιπόν ισχύει από τη γενική συζήτηση ως προς την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα αξιοπιστίας, δηλαδή οι αξιωματούχοι της Επιτροπής θα πρέπει να ε, εφαρμόσουν τις αποφάσεις που προκύπτουν από τη συναπόφαση τη δική σας και του Συμβουλίου. Όποια και να ήταν η πρόταση της Επιτροπής ε, έχει περάσει, παρήλθε. Ε, ψηφίσαμε να την εφαρμόσουμε. Και αν πείτε, α, η συναπόφαση ήταν ένα μεγάλο λάθος, τότε θα πρέπει να ανασταλεί η νομοθεσία, να αναπαιμφθεί και αυτό πρέπει να γίνει και αυτό με συναπόφαση. Δηλαδή, τι κάνετε, τηρείτε την νομοθεσία σας ή όχι. Και είναι δική σας η νομοθέτηση, δεν ήταν της Επιτροπής. Ήταν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Υπάρχει ένα τρίτο θέμα αξιοπιστίας. Ξέρετε ότι οι Αμερικανικοί αερομεταφορείς υπέβαλαν προσφυγή στο ΔΕΚ. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε γιατί είναι το ανώτατο νομοθετικό όργανο και είπε, αποφάνθηκε ότι συμβαδίζουν όλα με τους διεθνείς κανονισμούς και αυτούς που διέπουν τον ΙΚΑΟ. Έτσι αποφάνθηκε το ΔΕΚ. Σας, σας, σας τα υπενθυμίζω. Γιατί αν βάζετε ένα μεγάλο ερωτηματικό στην νομοθεσία, θα πρέπει να δείτε ποιος νομοθέτησε. Χρειάστηκαν δύο-τρία χρόνια συζητήσεων και εγώ ταξίδεψα ανά τον κόσμο εγώ ήμουνα ο πρώτος ε, ε, αξιωματούχος που αποτάνθηκε στην ΙΚΑΟ για παρόμοια θέματα και στην ΙΑΤΑ και ε, τότε είχαν όλοι ταχθεί υπέρ ενός συστήματος ε, αναγνώρισης εκπομπών και καταμέτρησής τους. Άρα αυτά δεν γίναν με σπουδή σαν να επρόκειτο για κάποιο διάταγμα της Επιτροπής το οποίο έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα. Το θέμα δεν αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο, διότι ο οικονομικός αντίκτυπος είναι περιορισμένος. Μιλάμε για λίγα ευρώ για μία πτήση μεταξύ Πεκίνου Φραγκφούρτης. Δεν πρόκειται για οικονομικό αντίκτυπο. Ξέρετε ότι αν και να αλλάξετε, ε, όταν αλλάξετε μία πτήση μέσω διαδικτύου, αν έχετε μία χειραποσκευή, θα πρέπει να καταβάλλετε πολύ περισσότερα από το κόστος αυτό που προαναφέρθηκε για τις εκπομπές. Πρόκειται όμως για ένα σύστημα αρχής, αρχών. Γι' αυτό θέλουμε να το αντιμετωπίσει η ΙΚΑΟ ως προς ε, την εξοεδαφική ερμηνεία. Εμείς έχουμε την υποστήριξη του ε, ΔΕΚ. Γι' αυτό μπορούμε να κοιτάξουμε οποιονδήποτε κατάματα. Πρόκειται για την εξοδικαστική φύση των εκπομπών του ETS. Και εδώ θα πρέπει να αποφανθούμε και γι' αυτό το συζητούμε εντός και εκτός ΙΚΑΟ. Όμως δεν μπορείτε να περιορίσετε την διεθνή αεροπλοεία στον εναέριο χώρο των κρατών, διότι πρόκειται για διεθνή χώρο αεροπλοείας και θα πρέπει να δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε, με, πώς θα αντιμετωπίσετε τις εκπομπές που δεν έχουν σχέση με τον κρατικό εναέριο χώρο. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία ελπίζω να επιλύσει ο ΙΚΑΟ. Ένα άλλο ζήτημα που μας απασχολεί και απασχολεί και την ΚΑΟ είναι η πρόσοδοι, διότι ε, τα, ε, οι πρόσοδοι είναι, αφορούν μάλλον ένα ε, θέμα καθαρά εκπομπών, αλλά το ζήτημα είναι πώς μπορούμε να φτάσουμε σε εισοδήματα κατά 15 ή 18% των εκπομπών που καλύπτονται από την αγορά αυτών των ποσοστώσεων. Όταν εγκρίθηκε το σύστημα με συναπόφαση, ελέγχθη ότι δεν ξέραμε πώς αυτά τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν, γιατί ένα κράτος μέλος θεωρούσε ότι τα κράτη-μέλη αυτόνομα θα αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα έσοδα. Και αυτό αντικατοπτρίστηκε στην τελική απόφαση. Άρα τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν. Εμείς έχουμε έναν μηχανισμό εποπτείας για να ρωτήσουμε τα κράτη-μέλη πώς δαπανούν ε, τις προσόδους αυτές. Η Γερμανία δημιούργησε ένα ταμείο όπου οι πρόσοδοι αυτοί από το ETS ε, μαζεύονται και πρόκειται για ποσά που πάνε στην έρευνα και στις υποανάπτυξη χώρες και πρόκειται για ποσά τα οποία ποτέ δεν θα φτάσει κανείς. Ως προς την εξοεδαφικότητα μπορούμε να το δούμε στα πλαίσια του ΙΚΑΟ και είμαστε, κρατάμε το κεφάλι ψηλά έτσι ώστε να μπούμε στις διαπραγματεύσεις με ψηλά το κεφάλι όπως είπα κάτι το οποίο δεν ακούσαμε εκτός ΙΚΑΟ. Γιατί ως προς το θέμα της αξιοπιστίας είδαμε ότι στη Μόσχα και, στο, στη Μόσχα και το ε, Νέο Δελχή μιλούσαμε εκτός ε, ΙΚΑΟ, δηλαδή να δούμε κατά πόσο θα υπερασπιστούμε τους οργανισμούς και τους φορείς ε, των Ηνωμένων Εθνών ή θα έχουμε ad hoc οργανισμούς όπως έγινε στη Μόσχα και στο Νεοδελχή. Αρκετά κράτη δεν ήταν παρόντα, δεν το θέλησαν γιατί δεν ήθελαν να ενθαρρύνουν ένα σκηνικό το οποίο θα αντιταχθεί του ΙΚΑΟ. Εκεί βρισκόμαστε σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο. Υπάρχουν δύο στοιχεία που σχετίζονται με, τη, με ενδεχόμενες αλλαγές. Ως προς τις εισερχόμενες πτήσεις υπάρχει μια διάταξη στην οδηγία του ETS όπου λέμε ότι οι ποσοστώσεις μπορούν να δοθούν υπέρ εκείνων που τις ζητούν και που καταδεικνύουν ότι έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα, μέτρα αντιστάθμισης δηλαδή. ποια είναι η αρχή που διέπει. Δηλαδή, αν μπορέσουμε να καλύψουμε τις εξερχόμενες πτήσεις, τότε καλύπτεται το θέμα με μία εισερχόμενη πτήση κάπου αλλού. Δηλαδή, ορίζουμε το ETS για τις εξερχόμενες πτήσεις, για τις αναχωρήσεις και αυτό αφορά τις αντίστοιχες αφήξεις. Έπρεπε λοιπόν να καλύψουμε τα μέτρα αντιστάθμισης, κάτι το οποίο έκανε ο νομοθέτης για εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις, αλλά δεν θελήσαμε να δώσουμε τελική μορφή στα μέτρα αντιστάθμισης, γιατί και ο ΙΚΑΟ θα διαδραματίσει ε, σημαντικό ρόλο. Ποια είναι, πώς έχει αυτή η αντιστήχηση θα πρέπει να το δει η διεθνής πολιτική αεροπορία. Μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε για τεχνολογία, για θέματα περιβάλλοντος, τεχνολογία και ασφάλεια. Εάν λοιπόν γίνουν συζητήσεις στον ΙΚΑΟ θα δούμε τι σημαίνει αυτή η αντιστήχηση, η αντιστάθμιση. Είναι δύσκολο να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει όμως να συγκρίνουμε ε, ε, μέτρα και όχι μόνο σε επίπεδο ETS. Εάν ο ΙΚΑΟ δεν βρει αντίστοιχα μέτρα για τις εισερχόμενες πτήσεις, τότε θα πρέπει να τροποποιήσουμε την νομοθεσία μας τα αντίστοιχα μέτρα για, την, ε, ε, για τις ερχόμενες πτήσεις μπορούν να επιληθούν μέσω επιτροπολογίας. Εάν όμως το ένα ή το άλλο στοιχείο δεν επιληθεί, τότε θα πρέπει να αλλάξουμε την ομοθεσία μας και να φτάσουμε στη συναπόφαση πάλι. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με σπουδή. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και αυτό το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Υπάρχει νομοθεσία μέσω συναπόφασης και μόνο μέσω συναπόφασης μπορεί να αλλάξει, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Τώρα, κατά πόσο υπάρχουν διαφορές στις συζητήσεις, τι γίνεται διεθνώς, τι βλέπουμε να κάνουν όλες οι χώρες οι οποίες αναφέρθηκαν. Ήπα, Κίνα, Ρωσία, Ινδία. Δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες, αλλά Γίνονται διμερείς συζητήσεις με όλες αυτές τις χώρες και βλέπουμε ότι υπάρχει στάση συνεργασίας από τις χώρες αυτές σε επίπεδο ΙΚΑΟ. Δεν λέω ότι όλες συμβαδίζουν, αλλά σας είπα ρητά ποια είναι η στάση τους και το γεγονός ότι θέλουν να συμβαδίσουν με τις ΙΠΑ γιατί η Ευρώπη και η ΕΠΑ έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, δηλαδή περίπου το 80% του παγκοσμίου μεριδίου το κατέχουν η ΕΠΑ και η Ευρώπη. Γι' αυτό προβάλλουμε μία ε, επιχειρησιακή συζήτηση, επιχειρησιακής φύσης συζήτηση με τις ΕΠΑ καταρχήν. Και υπάρχει πνεύμα συνεργασίας και από αυτές τις χώρες. Η Κίνα και η Ινδία έχουν περισσότερες αρχές ως προς τον εξοεδαφικό χαρακτήρα και τις προσόδους. Και εγώ επισκέφτηκα αυτές τις χώρες, ήρθα σε επαφή με τους ηθήνοντες και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε επίπεδο ΙΚΑΟ γιατί διαφορετικά μπορεί να έχουμε έναν ε, διτό χαρακτήρα διμερών επαφών, κάτι το οποίο δεν θα ήταν σκόπιμο για ε, θέματα αντιστήχησης και αντιστάθμισης. Τα δύο τελευταία ζητήματα. Τι θα γίνουμε αν υπάρξουν αντίπεινα. Από ό,τι βλέπω από τη δήλωση της Μόσχας, μιλάμε για ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς. Πρόκειται λοιπόν για ε, παράνομη διάκριση. Θα πρέπει όμως να διαφοροποιήσουμε για το τι λέγεται νόμιμα και επίσημα όταν γίνονται διασκέψεις ε, κορυφής και τι διαβάζουμε από τον τύπο πρόκειται για διαφορετικά ζητήματα. Ας θυμηθούμε ότι η Airbus ε, στην ουσία έχει εργοστάσια και στην Κίνα, τα οποία κατασκευάζονται εκεί. Κατασκευάζονται στην Κίνα, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες αυτές τις απειλές, δηλαδή ποιες είναι οι απειλές που ακούγονται στον τύπο και ποιες είναι οι επίσημες. Υπάρχει ο κίνδυνος αντιπίνων. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται, γιατί υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί. Και εάν υπάρχουν αντίτυπα κατά ενός εθνικού αερομεταφορέα υπάρχουν, υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει δυνατότητα προσφυγής και στο ΔΕΚ για να μην υπάρχουν διακρίσεις. Τέλος, πώς μπορούμε να, ε, τι μπορούμε να αντιτάξουμε και πώς μπορούμε να αποφύγουμε τον εμπορικό πόλεμο την εμπορική σύραξη. Γίνονται συζητήσεις στο ΝΙΚΑΟ. Και αν δεν είχαμε την νομοθεσία μας ETS, τότε δεν είχε καν αρχίσει η συζήτηση στον ΙΚΑΟ. Αυτό είναι το πρώτο σχέδιο. Το Plan A, που ε, αποτελεί την κινητήρια δύναμη του ΙΚΑΟ. Υπάρχουν ελπίδες ότι κάτι το πολύ θετικό θα βγει από όλα αυτά και μετά θα αποτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ε, πώς θα αποφανθεί ο ΙΚΑΟ και μετά θα γίνει μια άλλη συζήτηση. Και τότε θα πρέπει να αποτιμήσουμε την κατάσταση και να δούμε κατά πόσο ο Ευρωπαίος νομοθέτης βρίσκει τα στοιχεία αποδεκτά ή όχι. Για να αποφύγουμε λοιπόν την κλιμάκωση μία εμπορικής σύραξης, θα πρέπει να έχουμε μια καλή συνεργασία στον Νικάο και όπως είδαμε και στη δήλωση της Μόσχας και όπως ε, μας είπαν και από την Ινδία και από την Νότια Αφρική και από τις ΗΠΑ υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στο, στον Ότι έχουμε αυτή την ευκαιρία δεν έχουμε πολύ καιρό, αλλά εργαζόμαστε ως προς το πλάν A που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο προς το παρόν. Ελπίζω να υπάρχει και να γίνει μια καρποφόρα συζήτηση στον ΙΚΑΟ. Ευχαριστούμε κύριε Ντελμπέκ. Για την συνεισφορά σας και τις απαντήσεις σας. Ε, θέλω να, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε και άλλη συζήτηση. Είναι όντως διαδικαστικό ή είναι καμία ερώτηση. Ο κύριος Ντελμπέκε είπε αρκετά, αλλά δεν έμαθα τίποτα εγώ καινούριο. Κανένα σχόλιο όμως για το ζήτημα του ανταγωνισμού. Για το πώς ε, προκύπτει και τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Αν το εφαρμόσουμε εμείς και όχι οι τρίτες χώρες. Γιατί αυτό είναι θέμα ανταγωνισμού και δεν το αναφέρετε. Ναι, θα είμαι σύντομος. Όλα τα ζητήματα εφαρμογής καλύπτονται από τον νόμο ε, έχουν μέχρι σήμερα ακολουθηθεί ε, μητρώα δηλαδή παρακολούθηση και τα λοιπά όπως προβλέπεται από τον νόμο από όλες τις διεθνείς εταιρείες που πετάνε στην Ευρώπη σήμερα έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό θεωρώ εγώ. Και το λέμε και σε όλους τους διεθνείς εταίρους μας. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια κατάσταση αδύνατη για τις ε, αεροπορικές εταιρείες που θα πρέπει να διαλέξουν ε, σε ποια επικράτεια θα πάνε. Αυτό θα είναι το χειρότερο, διεθνέ, το χειρότερο αποτέλεσμα. Να πούμε δηλαδή σε αεροπορικέ εταιρείε και νομίζω το, το πείσαμε του Αμερικανού, γιατί ξέρετε και στη Γερουσία υπήρχαν κάποια νομοσχέδια που συζητούσαν και αν πείτε σε μια Αμερικανική εταιρεία είτε θα σεβαστεί τον Ευρωπαϊκό είτε τον Αμερικανικό νόμο ε, δεν, δεν συμβαίνει αυτό συνήθω στις διεθνείς επιχειρήσεις συνήθως σέβεσαι τον νόμο εκεί όπου δραστηριοποίησε. Και ήταν η Επίτροπος ξεκάθαρη, αν θέλει κανείς να λειτουργεί στην Ευρώπη, πρέπει να σέβεται τον Ευρωπαϊκό νόμο, όπως εμείς σεβόμαστε τους νόμους ε, άλλες χώρες όταν πηγαίνουμε και δραστηριοποιούμαστε εκεί. Είναι, ε, είναι ερώτηση ή διαδικασία. Άμα να ξαναξεκινήσει η συζήτηση, είναι ερώτηση γιατί ούτε τη δική μου ερώτηση η απάντηση. Τι θα γίνει με το φόρο στα αεροπορικά κάψιμα εάν... Ε, ε, δεν περάσει αυτό. Ναι, αυτό είναι, είναι ένα από τα στοιχεία που θα μπορούσα να είχα καλύψει στην ιστορική μου αναδρομή, γιατί ο φόρος στα αεροπορικά κάψιμα ήταν επιτάπητος σε πολλά κράτη-μέλη και χώρες ανά τον κόσμο και νομίζω πως πολλή στήριξη για το σύστημα αυτό υπήρξε γιατί προτιμούσαν μια διεθνή λύση εναρμονισμένη αντί για φορολογία που είναι μια εθνική υπόθεση τα, η φορολογία είναι εθνική όπως ξέρετε και και οι αεροπορικές εταιρείε συνειδητοποίησαν πως εάν σταματούσε αυτό το σύστημα θα είχαμε ξανά φορολογική προσέγγιση για τα καύσιμα, για τα εισιτήρια, για τα αεροδρόμια και ως καλύτερη λύση ε, προτίμησαν αυτό οι εταιρείε και όχι το, το άλλο σύστημα. Και μας το λένε Βεβαίω ε, μόνο ιδιωτικό, αλλά θα προτιμούσα να το λέγανε και δημοσίω. Αν δεν υπάρξει αυτό το μέτρο θα υπάρξουν φορολογικές ε, προσεγγίσεις ε, και πολύ εντονότερα όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη. Και μάλιστα υπάρχει κάποιο κράτος μέλος που είχε φόρους η Γερμανία και τους μείωσε για να αντισταθμίσει την εισαγωγή του συστήματο εμπορία εκπομπών που ξεκίνησε από πρώτης πρώτου. Απόδειξη λοιπόν του ότι αυτά ε, τα δύο συνδέονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντελμπέκε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να απαντήσετε σε ερωτήσεις μας. Και είμαστε γνώμονες, βεβαίως μας κρατάτε ε, ενήμερους για την πρόοδο που σημειώνεται. Ευχαριστώ πολύ. Okay, colleagues, we have one more item this... Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη σήμερα, σημαντικό. Ταμείο Συνοχής και κατάργηση του κανονισμού 1084 με κάποιες ειδικές διατάξεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση γνωμοδοτήσεις του κυρίου Κράμερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι ένα ευρύτατο έγγραφο που αφορά τους κανόνες οριζόντιους για όλα τα ταμεία. Και βεβαίως εμείς στην Επιτροπή μας βασιζόμαστε στα ταμεία συνοχής και τα περιφερειακά, γιατί εκεί πέρα ε, έχει σχέση η ε, συγκοινωνία, οι συγκοινωνίες. Ξεκινάμε με το Περιφερειακό Ταμείο. Ε, διατίθενται 376 δισεκατομμύρια. Τα 10 δισεκατομμύρια που θα πάνε για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από τα 376 είναι ψίχουλα. Και θέλω να παρατηρήσω πως υπάρχουν προβλήματα στη μετάφραση. Μα δεν ακούει. Ε, ήθελα να πω πως υπάρχουν προβλήματα στη μετάφραση γιατί στα αγγλικά μιλάνε ABCD στα γερμανικά ξεκινάνε από το B και όταν λένε άρθρο 7 στα γερμανικά είναι το 6 στα αγγλικά. Δηλαδή το σημείο B είναι στα γερμανικά, είναι εσύ στα αγγλικά. Ε, λίγο αστεία πράγματα. Προσέξτε το όμως. Ε, το προσέξαμε όταν διαβάζαμε τα έγγραφα. Λοιπόν, το άρθρο 3 ξεκάθαρα μιλάει για συγκοινωνίες, αλλά δεν μιλάει για βιώσιμες συγκοινωνίες. Και γνωρίζουμε πως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, σύμφωνα με την νομοθεσία τους στόχους 2020, πρέπει να προσανατολίσουν εκεί πέρα και θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές. Αυτό το έχει επιφασίσει και το Συμβούλιο. Οπότε θα πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις, οπότε θα πρέπει να μιλάμε για αηφόρες συγκοινωνίες και υπάρχει ε, έλλειψη της λέξης τουρισμού. Είμαστε Επιτροπή Μεταφορών, μεταφορών και Τουρισμού. Και η συνθήκη της Λισαβόνας επιτέλους και δικαίως ε, ε, έθεσε και τον τουρισμό υπό την αρμοδιότητά μας. Βεβαίω, το θέμα είναι και οι θέσει εργασία και κάναμε εμείς μια ανάλυση στο Περιφερειακό Ταμείο. 60% πάει στους δρόμους και μόνο 20% σιδηρόδρομου. οπότε οι επενδύσει δεν πάνε σωστή κατεύθυνση γιατί θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπέ και όχι να τι αυξήσουμε. Και ξέρουμε πώ οι οδικέ μεταφορέ είναι υπεύθυνε για το 72% των εκπομπών των μεταφορών. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να δώσω κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν πρέπει να επενδύουμε στη λάθος κατεύθυνση. λέμε πως καλό θα ήταν 40% ε, να πηγαίνει στον σιδηρόδρομο, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα κίνητρο και να λέμε, εάν παραδείγματο χάρη δίνονται 10 εκατομμύρια ε, στο σιδηρόδρομο και στα ποδήλατα, μπορούν να πάνε και 3 εκατομμύρια στις οδικές μεταφορές. Εάν πάνε 20 εκατομμύρια στα πρώτα που ανέφερα, μπορούν να πάνε πάλι ένα 30% στις οδικές μεταφορές. Οπότε να υπάρχει ένα κίνητρο να χρησιμοποιήσουμε τις ε, πιο φιλικές προς το περιβάλλον ε, μεταφορές. Μπορούμε ίσως να συμφωνήσουμε σε αυτό. Ένα σημαντικό βεβαίως θέμα είναι οι αστικές περιοχές και η αστική κινητικότητα. Ξέρουμε πώς είναι υπεύθυνε συγκοινωνίε για 30% των εκπομπών, αλλά στις πόλεις δεν είναι υπεύθυνε μόνο για 40% των εκπομπών, αλλά εάν δούμε όλες τις εκπομπές της πόλης, μιλάμε για ένα 70% των εκπομπών. Οπότε οι πόλεις έχουν μεγάλη σημασία, γι' αυτό η Κομισιόν έχει κάνει εκθέσεις για την αστική κινητικότητα, αλλά το πρόβλημα είναι πάντα η επικουρικότητα, γιατί κάποια μείνονται. Οι αστικές περιοχές είναι σημαντικές, ειδικά για τα λεφτά. Τώρα, αν επενδύσουμε στις δημόσιες ισοδιωτικές συγκοινωνίες, περισσότερα στις θέσεις εργασίας ε, χρησιμοποιούμε, ε, με συγχωρείτε, με τις δημόσιες, ε, τα δημόσια μας μεταφοράς. Αν δείτε π.χ. με την Ατλάντα με, στις, μία πόλη στην Ισπανία, η έκταση της Ατλάντας με μια πόλη δύο πληθυσμού στην Ευρώπη είναι 25 φορές μεγαλύτερη, είναι πολύ απλωμένη. Βεβαίως υπάρχει και υπο... το μετρό και οι υπόλοιπε, τα υπόλοιπα μέσα. Π.χ. το μετρό χρειάζεται μεγάλα μηχανήματα. Ε, στο δε Βερολίνο μπορούσαμε να κάνουμε ή 5 χιλιόμετρα μετρό ή 5, ε, ή ή 5 χιλιόμετρα μετρό ή 30 χιλιόμετρα τραμ. Δυστυχώ βέβαια η πόλη μου αποφάσισε για το μετρό. Αλλά θα πρέπει να μπορούμε να προωθήσουμε κάτι τέτοιο. Π.χ. στη Γερμανία έχουμε τον κανονισμό πως ε, ομοσπονδιακή χρηματοδότηση υπάρχει για το τραμ εάν ε, ε, έχουν μόνο δική τους ξεχωριστή λωρίδα τα τραμ. Π.χ. δεν θα υπήρχε στη Λισαβόνα τραμ γιατί οι γραμμές είναι μέσα στο δρόμο. Και γνωρίζουμε βεβαίως από την εμπειρία μας, είτε μιλάμε για την Κοπενχάγη είτε τη Σεβίλη, πως αν υπάρχει ε, τίτλος στον προϋπολογισμό για τα ποδήλατα επιταχύνεται πάρα πολύ η χρησιμοποίησή τους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα αηφόρο σχέδιο κινητικότητας και ανάλογη χρηματοδότηση για τα ποδήλατα. Στο άρθρο 7 το θέμα είναι ε, το ότι λείπουν ε, διάφορες συνδέσεις στην Ευρώπη, έχουμε πάρα πολλά κενά, το αναφέραμε, Πρέπει να γεμίσουμε αυτά τα κενά και να ασχοληθούμε και με το θόρυβο. Όλα αυτά μαζί ανήκουν στην ε, ευρωπαϊκή διάσταστα παραρτήματα. Πρέπει ε, να φροντίσουμε όχι μόνο να αυξάνονται οι αριθμοί των επιβατών, γιατί στα παραρτήματα αναφέρονται μόνο τα χιλιόμετρα. Καλό ακούγεται αυτό, αλλά η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με χιλιόμετρα σιδηροδρόμων. Αν δεν φροντίσουμε το υφιστάμενο δίκτυο, ε, δεν θα γίνει τίποτα. Πρέπει να δούμε όχι μόνο την ανάπτυξη του δικτύου, αλλά και την βελτίωση του, του υφιστάμενου. Και βεβαίως να μετατοπιστεί το δίκτυο από το δρόμο ε, στο σιδηρόδρομο και θα πρέπει στα αυτοκίνητα να βλέπουμε όχι μόνο την αύξηση των αυτοκινητοδρόμων αλλά και τη μείωση της κυκλοφορίας με αυτοκίνητο. Πάμε και μία εβδομάδα το μήνα στο Στρασβούργο, είδε κυρία Τροτμάν κατάφερε με με το τραμ να διώξει τα αυτοκίνητα από το κέντρο. Σας αναφέρω ένα παράδειγμα που το ξέρετε δηλαδή. Ε, τέτοια πράγματα πρέπει να σκεφτόμαστε. Όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Το ποσό είναι 68,7 δισεκατομμύρια ευρώ και θα πάνε πάλι 10 δισεκατομμύρια στα δύο ευρωπαϊκά δίκτυα. Οπότε 58,7 υπάρχουν, αλλά για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, συγκεκριμένα μέτρα βοήθειας δηλαδή. Και τα πράγματα τώρα είναι παρόμοια όπως και στο Περιφερειακό Ταμείο, δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά. Οι στόχοι του 2020 είναι σαφείς, ισχύουν και για το Ταμείο Συνοχής και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αυτό το οποίο λέμε, δηλαδή να αποφύγουμε ε, και να μετατοπίσουμε την ε, κυκλοφορία, γιατί μεταφέρονται πολλές βλακίες. Ορίστε. Και πολλές βλακίες λέγονται. Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ εγώ. Ε, auf jeden Fall, Ναι, ναι, βεβαίως, αναμένω να ακούσω και αυτά που θα πείτε. Οπότε μπορούμε να αποφύγουμε πάρα πολλά. Οι επενδύσεις λοιπόν πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια. Ε, δεν θέλουμε επενδύσεις που αυξάνουν, αυξάνουν τις εκπομπές. Δεν θέλουμε επενδύσεις που μειώνουν την ευρωπαϊκή προστασία αξία. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Δεν θέλουμε εκπομπές που επιβαλύνουν το περιβάλλον στο μέλλον και να το πληρώνουν τα παιδιά μας. Ε, είτε μιλάμε για οικονομικές ζημιές είτε για περιβαλλοντικές. Και δεν θέλουμε επενδύσεις που αυξάνουν το εξωτερικό κόστος. Το παράρτημα και στο Ταμείο Συνοχής είναι παρόμοιο με το, Περιφερειακό Ταμείο. Αυτά λοιπόν ως πρώτη παρουσίαση. Αναμένω τώρα τις ε, φορές των συναδέλφων και μετά θα μπούμε πιο συγκεκριμένα στο θέμα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας. Γκρός e. για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Κράμερ για την εισαγωγή. Αυτό το οποίο προτείνει εδώ πέρα η Κομισιόν, αν το συγκρίνουμε με το παρελθόν για τα διαπτωτικά ταμεία, είναι πολύ ενδιαφέρον, ειδικά για εμάς, στην Επιτροπή μας. Θεωρώ πως το έχει είναι στόχοι με τους οποίους συμφωνούμε όλοι, είτε μιλάμε για το 2020, κοινωνικές, οικονομικές στοιχές, αηφορία. Που υπάρχει πάρα πολύ, σε πάρα πολλά κεφάλαια, για αηφορία μιλάει και περιβάλλον. Αλλά θεωρώ πως θα πρέπει εδώ πέρα να εκμεταλλευτούμε την ε, ευκαιρία αυτό το οποίο η Κομισιόν ε, ονομάζει ερεσιμότητα, να το τονίσουμε περισσότερο. Να επανέλθω όμως στη χρηματοδότηση. Όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, πρέπει εδώ πέρα στην έκθεση να υπάρχει βεβαίως η σύνδεση με το, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, αλλά και το νέο μέσο χρηματοδότησης, το οποίο αναφέρεται και ε, τα ομόλογα έργου, να γίνει δηλαδή πιο ξεκάθαρο και να μπορέσουμε να πούμε σε ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει κάτι τέτοιο δεύτερον. Σημαντικό είναι εμείς εδώ στην Επιτροπή να ξεκαθαρίσουμε πως οι επενδύσεις στις μεταφορές είναι διπλά θετικές και να μην υπάρχει η ε, πεποίθηση πως παίρνουμε εμεί λεφτά από το Ταμείο Συνοχής. Τα λεφτά ούτως ή άλλως θα πήγαιναν για την κινητικότητα και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε ε, την ευκαιρία να καθησυχάσουμε δηλαδή και να λέμε πως ούτως ή άλλως εκεί θα πήγαιναν τα λεφτά. Τώρα, για την... Ε, για την αιρεσιμότητα αυτή. Υπάρχει, όπως ξέρετε, το υλικό και το λογισμικό θα έλεγε κανείς στις ε, μεταφορές ε, και αυτό το οποίο συζητάμε τους ε, τελευταίους μήνες. Και πράγματι δίκαιο έχετε, έχουν ξεχάσει τον τουρισμό, πρέπει να τον αναφέρουμε περισσότερο στα διάφορα προγρήματα. Το γεγονός πως και εδώ πέρα θα πρέπει να αναφέρουμε το διοξίδιο του άνθρακα και μπορούν νομίζω έτσι να αναφερθούν οι μεταφορές. Οι γέφυρες με τα διευρωπαϊκά δίκτυα με το βασικό και το εκτεταμένο δίκτυο όπου θεωρούμε πως θα πρέπει να υπάρχει μια συμπληρωματικότητα και τα διαρθρωτικά ταμεία να χρησιμοποιηθούν και στις ε, τοπικές επενδύσεις για να μπουν σε ένα συνολικό πλαίσιο. Αυτό νομίζω είναι μια πραγματική Τα Αυτό το οποίο επίσης δεν αναφέρεται αρκετά είναι το κοινωνικό ταμείο και ειδικότερα οι δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Εάν βλέπετε πως υπάρχει ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό. Μπορούμε να δώσουμε λοιπόν έμφαση σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά τις μεταφορές και τη γεννητικότητα. Η νέα αρχή ή η ενισχυμένη αρχή της εταιρικής σχέσης είναι επίσης σημαντικό για μένα γιατί γνωρίζουμε ήδη πως υπάρχουν χώρες που θέτουν ερωτήματα για τη χρήση των διευρωπαϊκών δικτύων και για το εάν εξακολουθεί να υπάρχει κάποια επικουρικότητα. Οπότε η εταιρική αυτή σχέση, όπου μιλάμε από τους μικρούς μέχρι τους μεγάλους, νομίζω είναι ένα κομμάτι της απάντησης σε αυτή την ερώτηση για το εάν το τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο χρησιμοποιείται ή εάν υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία υπαγορεύονται Οπότε νομίζω έτσι μπορούμε να έχουμε ένα έργο το οποίο αναπτύσσεται τοπικά με συγκεκριμένα κριτήρια και συνεχίζει. Οπότε για μένα αυτό είναι μια σημαντική ε, απάντηση. Όσον αφορά δε τα οικονομικά μέσα και την επικουρικότητα πρέπει να το τονίσουμε. Τώρα σύγχρονες τεχνολογίες είτε μιλάμε για πληροφορική επικοινωνίες θα μπορούσαν να αφαιρθούν πολύ περισσότερο και τελευταία πτυχή και αυτό αφορά και αυτό το οποίο είπαμε στις μεταφορές να μην αναφέρουμε μόνο ότι υπάρχουν στενοποί αλλά να υπάρχει δυνατότητα επένδυσης. Χτες είπε ένα συνάδελφος πως τα διευρωπαϊκά δίκτυα δεν, είναι, δεν έχουν στόχο να ενώσουν δύο χωριουδάκια αλλά τα μία θα μπορούσαν να δράσουν συμπληρωματικά ε, για τέτοιες υποδομές. Αυτά είναι νομίζω πράγματα που θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε για τις μεταφορές, κινητικότητα, τουρισμό κτλ. Για να δώσουμε απαντήσεις σε ερωτήσεις που θα μας ε, απασχολήσουν. Για τη χρήση των, ταμείων, των κονδυλίων στο Ταμείο Συνοχής. Ευχαριστώ, eh, eh, Σενάλοβα. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω κάνοντας κάποιες γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ταμεία Είμαι σαφώς υπέρ της πρότασης γιατί έχει ως στόχο να πετύχει ένα υψηλότερο επίπεδο ελέγχου, θέτει συγκεκριμένου στόχους και προτείνει ένα καλύτερο σύστημα χρηματοδότησης ορισμένων έργων. Όσον αφορά τις μεταφορές, θα ήθελα να φερθώ στην στρατηγική προτεραιότητα παριθμών 7. Είμαι σαφώ υπέρ των βιώσιμων μεταφορών και την απομάκρυνση στενοπών σε κάποιες πολύ σημαντικές υποδομές. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών, κυρίως στα νέα κράτη-μέλη. Στα νέα κράτη-μέλη πρέπει να έχουμε και ευρία δίκτυα μεταφορών, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε μια καλύτερη εδαφική συνοχή. Αποδεχθήκαμε, όπως ξέρετε, αυτό, το, το στόχο στη Λευκή Βίβλο Μεταφορών και πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2015. Σαφώς θα πρέπει να υποστηρίξουμε και τις βιώσιμες μορφές μεταφορών. Πρέπει όμως να γίνει περισσότερη συζήτηση για συγκεκριμένα ζητήματα ιδίως για τον προπολογισμό τα 10 δισεκατομμύρια για τις ε, διασυνδέσεις στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε κάποιους ξεκάθαρους κανόνες για το πώς τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να προτιμάσουν κάποια έργα και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν και την επαρκή χρηματοδότηση. Τώρα, η αρχή της αλληλεγγύης δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υποκατασταθεί από την αρχή του ανταγωνισμού ανάμεσα σε κράτη-μέλη του Ταμείου Συνοχής. Ο κύριος Γκρός αναφέρθηκε συμφωνία όσον αφορά την εταιρική σχέση με σαφώς υπέρ των εταιρικών σχέσεων, γιατί πιστεύω ότι συμπεριλαμβάνουν πολύ περισσότερο το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο και δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στις τοπικές ανάγκες. Ένα ζήτημα το οποίο θέλω να συζητήσουμε περισσότερο στο μέλλον είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων βάσει συγκεκριμένων δικτών. Για παράδειγμα, όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Οι συνάδελφοι επίσης αναφέρθηκαν στην μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Η αιρεσιμότητα αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να δίνει τα απαραίτητα κίνητρα στα κράτη-μέλη για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους, για να εναρμονίσουν τελικά τους στόχους τους με τις ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσε να θέσει κανείς ένα αμφιβόλο αν όντως η αιρεσιμότητα θα πρέπει να πάρει αυτή τη μορφή. Νομίζω ότι η αιρεσιμότητα θα πρέπει να συνάδει με στόχους της πολιτικής συνοχής. Ένα εξίσου σημαντικό σημείο είναι το απόθεμα 5% από το Ταμείο Συνοχής που θα δοθεί στα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία έχουν πετύχει συγκεκριμένα επιτεύγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τόσο τον θετικό όσο και τον αρνητικό αντίκτυπο μιας τέτοιας πρότασης. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για το Ταμείο Συνοχής. Επομένως θα ήθελα και προς αυτό να κάνω κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Βλέπουμε ότι η πρόταση αυτή προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ωστόσο πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο. Όπως και χθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα Ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στην υφιστάμενη υποδομή των κρατών μελών και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρους ορισμούς και ξεκάθαρους δείκτες για την προετοιμασία των έργων. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε επίσης μετρήσιμα αποτελέσματα και συγκεκριμένους δείκτες για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης όσον αφορά τα επιτυχή έργα. Είμαι επίσης υπέρ των προσπαθειών που γίνονται για να μειωθεί η γραφειοκρατία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε επίσης και πιο σημαντικούς ελέγχους όσον αφορά την χρήση των ταμείων αυτών. Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε κράτη-μέλη του Ταμείου Συνοχής. Επίσης γίνεται και μία συζήτηση όσον αφορά τη μεταφορά αυτών των 10 δισεκατομμυρίων, το οποίο φτάνει τελικά το 15% της χρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής. Πρέπει να έχουμε σαφείς όρους έτσι ώστε να μην χαθεί η χρηματοδότηση για κάποια σημαντικά έργα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα έργα θα τυχαίνουν ενό πολύ καλού συντονισμού από τους Ευρωπαίους συντονιστές. Πρέπει να έχουμε επίσης ένα σαφή ορισμό για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επίσης θα πρέπει να να διευκρινίσουμε, να εντοπίσουμε κάποιες ανάγκες όσον αφορά τα έργα τα οποία υπάγονται στο CEF, το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Επίσης, η κατανομή των πόρων για τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να μειωθεί. Η αρχή use it or lose it από όλες σε περίπτωση μη χρήσης είναι πολύ σημαντική ως προς αυτό. Όσον αφορά τώρα τα ανώτατα όρια, 2,5% του ΑΕΠ, Καταλαβαίνω σαφώς εδώ πέρα τις προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου να επιτευχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς μειώντας απλώς τα εγκεκριμένα έργα. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξορθολογήσουμε καλύτερα την πραγματοποίηση των έργων και να μειώσουμε το διοικητικό άχθος. Επίσης θα πρέπει να σας απασχολήσει και η γενικότερη επίπτωση αυτού του κανονισμού. Και αυτό το 2,5% του ΑΕΠ. Και μια τελευταία παρατήρηση όταν θα επιλέγουμε τις επενδυτικές προτεραιότητες, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις ασφαλείς υποδομές. Νομίζω ότι οι ασφαλείς οδικές υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Πάνω από το 75% των οδικών ατυχημάτων γίνονται σε μικρούς επαρχιακούς δρόμους. Επομένως η ασφάλεια στους δρόμους, η ασφάλεια στο δικό δίκτυο είναι μια πολύ σημαντική προτεραιότητα στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές ε, θέτουμε μία ημερομηνία η οποία φτάνει μέχρι το 2015. Νομίζω ότι κάποιοι άλλοι στόχοι φτάνουν μέχρι το 2020, αυτές οι ημερομηνίες που έχουμε. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κράμερ για την παρουσίαση που έκανε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε κάποια βασικά σημεία προτού καταλήξουμε στο σχέδιο έκθεσης. Εργάζομαι επίσης και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και θα ασχοληθώ και στην Επιτροπή αυτή με το ζήτημα αυτό το οποίο εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Νομίζω λοιπόν ότι Το έγγραφο αυτό είναι πολύ καλό και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν κοινό κανονισμό και για, τα, για όλα τα ταμεία. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε και εμείς προσπάθειες προκειμένου να καταφέρουμε να συγκεράσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές πολιτικές σε μια κοινή προσέγγιση, να έχουμε έναν ε, εξορθολογισμό όσον αφορά την ε, κατάρτιση του κανονισμού αυτού. Νομίζω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε λοιπόν την ε, γνώμη μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τις αμφιβολίες που έχουμε όσον αφορά τον αποκλεισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την κοινή στρατηγική νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με αρκετό σθένος και να πούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει και εμείς να ανήκουμε στην όλη διαδικασία του διαλόγου, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Δεν μπορούμε να μείνουμε στο περιθώριο και να αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο μόνο να κάνουν όλη την ουσιαστική εργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα και να τοποθετηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει την εργασία της από την δική της την πλευρά, στην κατάρτιση δηλαδή των προτεραιοτήτων της. Εναπόκειται λοιπόν τώρα σε εμά να κάνουμε τη δική μας την εργασία και να δώσουμε εμεί κάποιε συγκεκριμένε ενδείξεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σωστά ορισμένοι συνάδελφοι εξέφρασαν κάποιες ανησυχίες και κάποιες αμφιβολίες. όσον αφορά τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των μεταφορών, προφανώς αναφερόμαστε στις βιώσιμες μεταφορές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε όσον αφορά το σημείο αυτό. Το έχουμε λοιπόν συνεχώς κατά νου. Ένα άλλο σημαντικό κεφάλαιο έχει να κάνει με την αιρεσιμότητα ex ante και ex post. Νομίζω ότι θα πρέπει η αιρεσιμότητα να ισχύει εκ των προτέρων περισσότερο, δηλαδή εξ αρχής να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι όροι ρυθμίζουν ουσιαστικά την κατανομή των πόρων. Τι θα πρέπει δηλαδή γενικότερα να ισχύει όταν δεν εντοπίζεται κάποια παραβίαση των κανόνων. Δηλαδή, ποιε είναι οι κατευθυντήριε γραμμέ που θα πρέπει να ακολουθούν οι περιφέρειες στην έγκριση συγκεκριμένων έργων. Τώρα, πώς έχει κατάσταση εξπόστα εκ των υστέρων. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί να σας πω καταρχάς ότι έχουμε μία και μοναδική συγκεκριμένη σύμβαση εταιρικής σχέσης και έχουμε πολλές διαφορετικές περιφέρειες στη συνέχεια. Ορισμένες λειτουργούν σωστά και κατανέμουν σωστά τους πόρους, ενώ έχουμε και άλλες περιφέρειες από την άλλη που δεν είναι τόσο ενάρετες θα έλεγα. Δεν μπορούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε μία κοινή μοναδική λύση για όλους. Θα πρέπει αυτό να μας απασχολήσει και δεν θα πρέπει να παραχωρήσουμε μία επιταγή ελευκό. Προχωράει πάντως ε, ο χρόνος να κάνω μία ακόμα τελευταία παρατήρηση. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν για την νομοθετική δέσμη για τους σιδηροδρόμους και για την σχετική αιρεσιμότητα που θα πρέπει να ισχύει. Για άλλη μια φορά πάντως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να αναφερθούμε ξεκάθαρα και στον τομέα του τουρισμού και ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τον πολύ σημαντικό αυτό κλάδο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ρικέ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Μάικλ Κράμερ για την παρουσίαση που έκανε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, αναφερόμαστε εδώ πέρα σε έναν χρηματοοικονομικό κανονισμό. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για το κείμενο αυτό. Και θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να ερμηνεύσουμε και το κείμενο. Δεύτερον, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα διαρθρωτικά ταμεία όπως το ΦΕΝΤΕΡ για παράδειγμα και το Ταμείο Συνοχής. Τα διαρθρωτικά ταμεία ΦΕΝΤΕΡ είναι ταμεία τα οποία εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο Δηλαδή, προηγείται ένας διάλογος ανάμεσα στο κράτος μέλος και την περιφέρεια, ενώ το Ταμείο Συνοχής υφίσταται σε εθνικό επίπεδο και εκεί πέρα εφαρμόζεται η χρηματοδότηση. Και αυτό επηράζει τα πράγματα όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Οι ε, δικές μας, τα, τα σχέδια τα οποία εμείς προωθούμε είναι περισσότερο θεματικά σχέδια, διασωνοριακά θέματα, αυτά τα οποία εντάσσονται ουσιαστικά στην Ευρώπη 2020. Προωθούμε ουσιαστικά την εφαρμογή έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε εξ αρχής. Να επενθυμίσω επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Τα, ταμεία που δίνονται, τα που δίνονται για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών είναι κυρίως περιφερειακή Ακόμα και για μεταφορές ουσιαστικά διασυνοριακές έχουμε περίπου 27 δισεκατομμύρια που δίνονται μέσω των περιφερειακών ταμείων. Για να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο εκτελεστικός προπολογισμό που υπάρχει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, που πολλές φορές μιλάμε για το 1 δισεκατομμύριο, βλέπουμε τελικά ότι περισσότεροι πόροι θα πρέπει να έρθουν από τα περιφερειακά ταμεία. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης εξάντε. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει είτε για κάποιες θεματικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως αυτή, είτε γενικότερα για τα έργα της Στρατηγικής Ευρώπη 2020. να πω κάποια πράγματα όσον αφορά τα ταμεία συνοχής, όχι μόνο επειδή είμαι σκιώδης ηγητής, αλλά επειδή μας ενδιαφέρει και το ταμείο αυτό πολύ περισσότερο στα πλαίσια του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη. Το μέσο αυτό προτείνεται να έχει 67 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια αρχική πρόταση στα πλαίσια της συζήτησης που θα γίνει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτά τα 67 λοιπόν δισεκατομμύρια θα πάνε προς έργα μεταφορών, θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία καλύτερων περιβαλλοντικών συνθήκων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος του ποσού αυτού δίνεται για τις μεταφορές. Κάτι το οποίο δεν αναφέρεται και αποτελεί πρόβλημα αυτό για μας είναι ότι δεν δίνονται συγκεκριμένες ενδείξεις ως προς τα έργα μεταφορών που θα μπορούσαμε να προωθήσουμε. Τα πράγματα στην καλύτερη περίπτωση είναι πάρα πολύ ασαφή στην πρόταση κανονισμού. Για παράδειγμα, θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη ε, σημασία στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, στην διατροπικότητα, στο πόσο εγκάρσια οριζόντια μπορεί να είναι τα σχέδια αυτά. Στα ζητήματα αυτά η πρόταση αναφέρεται πολύ λίγο. Και υπάρχει και ένα ακόμα σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει πολύ. Ποιο θα είναι το ποσό το οποίο θα δοθεί σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Θα γίνει μία εκ των προτέρων κατανομή των πόρων. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική συζήτηση που γίνεται τώρα στο Συμβούλιο και τα ποσά τα οποία θα δούνε θα πάρουν τη μορφή επιχορηγήσεων, θα πάρουν τη μορφή κάποιων εγγύσεων. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι ποσοστό κοινοτικών κονδυλίων θα μπορούσε να δοθεί στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα επιλεγούν τελικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί. Τώρα, η αρχή του θα, ότι εξυπηρετείται αυτός ο οποίος φτάνει πρώτος, αυτός που κάνει το αίτημα πρώτος, είναι μια αρχή η οποία προκαλεί πολλά προβλήματα σε ορισμένες χώρες. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν στα πλαίσια ενός δημοσιονομικού κανονισμού να καταφέρουμε να διαχειριστούμε ζητήματα όπως η κατανομή των πόρων και η διαχείριση των πόρων αυτών. Επίσης, το, ο, ο εγκάρσιος χαρακτήρας, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει στα έργα στα οποία αναφερόμαστε εδώ πέρα και όπως είπε και ο Μάικλ, είναι καλύτερο να αναφερθούμε στα έργα αυτά τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένο αριθμό χιλιόμετρων ανά επιβάτη. Επίσης, Γίνεται κάποια, ε, προτείνονται κάποια έργα τα οποία εντάσσονται στα European Facilities, 10 δισεκατομμύρια. Η κατανομή θα γίνει από, την, από τον εκτελεκτικό, εκτελεστικό με οργανισμό. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ε, πώς ακριβώς θα γίνει η κατανομή των σχετικών αυτών πόρων. Τα πράγματα μένουν πάρα πολύ ασαφή σε πάρα πολλά σημεία όσον αφορά αυτή την πρόταση κανονισμού. Η κυρία Τσικάου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κράμερ για την παρουσίαση. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε και τις εκθέσεις. Θα ήθελα να κάνω μία γενική παρατήρηση. Όταν μιλούσαμε για μία οδηγία για, την για τις ελλείψεις μάλλον στον ε, τομέα ενέργειας στην Ήτρε μιλούσαμε για θέματα που άπτονται των διαρθρωτικών ταμείων. Μας είχαν πει λοιπόν τότε ότι το έγγραφο πλαίσιο δεν είναι νομοθετικού χαρακτήρα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, σημεία αναφοράς. Ελπίζω να μην συμβεί ε, αυτό και με το συγκεκριμένο πακέτο, δηλαδή να υπάρχει νομοθετική συνοχή όλα τα βασικά στοιχεία που είναι οι περιορισμοί ή η εκλογιμότητα να προβλέπονται στον κανονισμό και όχι σε άλλα κείμενα στα οποία να αναφερόμαστε όπως ε, μάλλον ενίδη γενικού πλαισίου να υπάρχει δηλαδή ε, νομοθετικό περιεχόμενο ως προς τις αστικές μεταφορές νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας αυτό το θέμα, δηλαδή να ενταχθεί στους κανονισμούς περί διαρθρωτικών ταμείων. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή, όπως είπε ο κύριος Ρίκε, ότι υπάρχουν ταμεία που αφορούν και την περιφερειακή ανάπτυξη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την επικουρικότητα. Θυμίζω ότι στον στη Λευκή Βίβλο που εγκρίναμε πέρσι γίνεται λόγος για αστικές μεταφορές. Θα πρέπει δηλαδή στο επόμενο πολιετές πλαίσιο να χορηγούνται κονδύλια μόνο όταν υπάρχει ένα σχέδιο ανάπτυξης ε, αστικών μεταφορών και ένας εξωτερικός αυτόνομος έλεγχος, ο οποίος να πιστοποιεί αυτό το σχέδιο ή πρόγραμμα. Γιατί ελοχεύουν πολλοί κίνδυνοι και υπάρχουν και αντιφάσεις ως προς την αρχή της επικουρικότητας. Ελπίζω το θέμα αυτό να διασαφινιστεί μέσω κανονισμών, τους οποίους συζητούμε, ως προς την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για το, και για τα 10 δις από το Ταμείο Συνοχής. Πιστεύω ότι αυτά τα κονδύλια να ε, αφορούν τις ε, περιφέρειες για, ε, που εντάσσονται στο στόχο σύγκλησης για τις αστικές μεταφορές. Στο χρηματοδοτικό πακέτο για το μελλοντικό πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη χάνουν 10% από τα διαρθρωτικά ταμεία και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα δέκα δις ε, που θα αφορούν τις μεταφορές, που θα εγγραφούν για τις μεταφορές για τα νέα κράτη-μέλη υπό το στόχο της σύγκλησης, να μην θεωρηθούν χαθούν κονδύλια που θα χαθούν για αυτά τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ε, θα ήθελα να αναφερθούμε στην εθνική κατανομή για τον τομέα των μεταφορών, γιατί υπάρχει μεγάλο έλλειμμα για τις ε, μεταφορές στις νέες χώρες. Αυτό αφορά και τις σιδηροδρομικές και την αυσιπλοεία αλλά ε, στα νέα κράτη-μέλη υπάρχουν πολύ υψηλές ανάγκες και για τις οδικές μεταφόρες. Αν ε, για τη Γερμανία είναι οι οδικές μεταφορές ε, μολύνουν το περιβάλλον, μπορώ να σας πω ότι στη Ρουμανία μολύνουν πολύ περισσότερο οι οδικές μεταφορές. Γι' αυτό θα πρέπει να μας υποστηρίξετε για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, για την διατροπικότητα, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες ανάπτυξης των υποδομών μεταφορών στα νέα κράτη-μέλη. Και ελπίζω αυτό να ενταχθεί και στους νέους κανονισμούς που αφορούν τις μεταφορές. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που θίξατε. Η αρχή χρησιμοποίησε το ή χάσε το, το use it or lose it. Εάν λάβουμε υπόψη την χρηματοοικονομική κρίση υπάρχουν επιπτώσεις ανάλογα με τη χώρα για την οποία μιλάμε. Θα πρέπει να ληφθεί όμως πολύ σοβαρά αυτή η αρχή του use it or lose it, γιατί υπάρχει μεγάλη ε, χρηματοοικονομική πίεση για ορισμένα κράτη και δεν μπορούν να κινηθούν με την ίδια σπουδή. Γιατί ε, αρχηγός, αρχικός είχαν γίνει άλλες προβλέψεις και μετά άλλα κράτη ε, αποδείχθηκε πως ήταν υπερχρεωμένα. Οπότε θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με ορισμένα κράτη ε, με την αρχή αυτή άμα τα αφήσει ε, σαφήνει, ειδικά για τις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση. Δεύτερον, η κυρία Τικάου το ανέφερε. Ναι, βεβαίως, κάποιες από τις νέες χώρες υπάρχουν ε, κάποια προβλήματα, π.χ δεν υπάρχει παραδείγματο χάρη σε μια γειτονική χώρα ή ανάλογη υποδομή. Αλλά βεβαίω θα πρέπει να πούμε πω εάν παίρνουμε σοβαρά την αρχή της αηφορία, δεν θα πρέπει οπωσδήποτε όλα τα λάθη τα οποία κάναμε στην ε, Δυτική Ευρώπη να τα επαναλάβουμε και στα νέα ε, Έχουμε πολλές εμπειρίες για το ότι δεν δημιουργεί κάθε υποδομή λύση των προβλημάτων της συγκοινωνίας. Αντιθέτως, καμιά φορά τα επιδεινώνει. Γι' αυτό, κατά την άποψή μου, ακριβώς η αρχή που αναφέρθηκε με το ΕΞΑΝΤΗ και το εξπόστ, τους ελέγχους αυτούς, ε, νομίζω είναι βασική. Στην Επιτροπή Δενομικών Υποθέσεων ε, ασχολούμαι με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και είναι πολύ ε, απογοητευτική κατάσταση πως ε, διαπιστώνουμε πάντα εκ των υστέρων πως είχαμε ε, λάθη και δεν ανταποκρινόμασταν στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προειδοποιείται το χύψη ε, κράτος μέλος και αυτό οδηγεί στη διόνυση λαθών και δεν λαμβάνεται υπόψη το τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού και αυτοί οι οποίοι κάνουν ε, αυτά τα λάθη ε, αποφασίζουν από κοινού για επενδύσεις στις ευρωπαϊκές υποδομές. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα το οποίο έχουμε πάντα. Και παραδείγματο χάρη ειδικά όσον αφορά τις οδικές μεταφορές θα πρέπει να έχουμε κάποιες προβλέψεις εξ άντε. Μια εταιρική σχέση την οποία ε, δηλώνουμε και μετά βλέπουμε πως δηλώνονταν μόνο προϊόντα τα οποία σταδιακά δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια θα είναι κάτι το πολύ περίεργο. Δηλαδή εκεί πέρα γνωρίζω πως ε, πολλά νέα αλλά και παλαιά ε, θέλουν να αποφασίζουν μόνα τους και ε, το τι θα πρέπει να κατασκευάζετε, αλλά το ζήτημα είναι το τι θα πρέπει να, χρημα... να συγχρηματοδοτείτε. Εάν εκεί ε, σιγά σιγά απομακρυνθούμε από τις αρχές τις οποίες ε, έχουμε, ε, γιατί μιλάμε για τεράστια κλίμα, ε, τεράστια χρήματα, θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την αξιοπιστία και τις αρχές μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι αρχές. Οπότε για μένα το ερώτημα είναι εάν είναι ρεαλιστική μια τέτοια εταιρική σχέση όταν οι προθέσεις κάποιων κρατών μελών πηγαίνουν σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Τέλος η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή τον εισηγητή, τον κύριο Κράμερ και θα ήθελα να τονίσω ορισμένες πτυχές. Να δούμε δηλαδή πού θα γίνουν οι μεγαλύτερες επενδύσεις από τον προϋπολογισμό και μας ενδιαφέρει και η πράσινη εργασία, δηλαδή οι θέσεις εργασίας που αφορούν την ανανεώσιμη, την βιώσιμη, με συγχωρείτε, ανάπτυξη και την πράσινη ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να μας πει η Κομισιόν κατά πόσο έχει επαρκή αριθμητικά στοιχεία για να μπορέσει να αναλύσει αυτή την προστιθέμενη αξία εάν υφίσταται και επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα των βιώσιμων μεταφορών. Όπως ήδη είπαμε σε ορισμένα κείμενα, πέρα από την τοπική συνεργασία και όλη τη στρατηγική συνεργασίας, υπό εθνική επιτήρηση, θα πρέπει να γίνει λόγος και για ένα επίπεδο επίλυσης διαφορών. Όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλες υποδομές ή σημαντικές επενδύσεις, όπου υπάρχει συναπόφαση σε ευρωπαϊκό και κρατικό επίπεδο, για να ξέρουμε τι ε, συνέργεια χρειάζεται μεταξύ δημόσιου, κρατικού τομέα και ευρωπαϊκού. μέσα στα πλαίσια και των εθνικών στρατηγικών για την ανάπτυξη των υποδομών. Γιατί πολλές φορές φαίνεται ότι πρόκειται για αποφάσεις εκ των άνω που πέφτουν στο τοπικό επίπεδο και οι τοπικές αρχές δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτές τις αποφάσεις ή τα προγράμματα. Θα πρέπει λοιπόν και οι Κομισιό να μας υποστηρίξει, διότι φαίνεται να ύπταται αυτή η περίφημη επικουρικότητα, χωρίς να ξέρουμε πώς ακριβώς θα ενσωματωθεί στον ε, ιστό των αστικών μεταφορών. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε και τον τουρισμό, ο οποίος ε, ε, αποτελεί κινητήριο δύναμη. Θα πρέπει να υπάρχει νομική βάση και συγκεκριμένη στρατηγική, γιατί για πρώτη φορά στα πλαίσια της ευρωπαϊκής εδαφικότητας λαμβάνουμε υπόψη περιφέρειες που εντάσσονται ή που ενδεχομένως δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο, γιατί μιλάμε και για όμορες περιοχές. Ε, ο κύριος Κράμερ είπε ότι για πρώτη φορά υπάρχουν ε, και υπάρχει και το μαστίγιο αλλά και το καρότο από, στιγμή από σημείο σε σημείο, κάτι το οποίο δεν υπήρχε μέχρι του δεν Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό και στις κατεξουσιοδότηση πράξεις, δηλαδή στα πλαίσια του μαστιγίου και του καρότου, να ενισχύσουμε το σκέλος του καρότου. Επιτροπή, κυρία Λανχάιερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και όλους αυτούς που πήραν το λόγο και κάλυψαν πάρα πολλά ζητήματα. Θα ήθελα να φερθώ σε κάποια από αυτά απαντώντας κι εγώ τα όσα υπόθηκαν στις παρεμβάσει αυτές έχουν να κάνουν με τα όσα προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε με το σχέδιο νομοθετικής πρότασης. Καταρχάς, να επικεντρωθούμε στην Ευρώπη 2020. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα προγράμματα χρηματοδότηση, όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότηση θα επικεντρωθούν στο να επιτευχθεί ο στόχο τη εφιούς βιώσιμη ανάπτυξη. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε στα πλαίσια τη πρόταση αυτή να συγκεράσουμε και τα πέντε αυτά ταμεία και να καταφέρουμε μέσω τη εταιρική σχέσης να χρηματοδοτήσουμε συγκεκριμένα έργα στη συνέχεια. Όσον αφορά το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, αναφέρθηκε σε ορισμένε παρεμβάσει αυτό. Όπω υπόθηκε, προτείνουμε να γίνει μέσω κατεξοδότηση πράξη, δηλαδή όπω όπως επιτρέπει και η νέα συνθήκη. Υπάρχουν όμως και κάποια ερωτήματα στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει αυτή τη στιγμή, τις επόμενες ημέρες, ένα έγγραφο το οποίο θα δίνει περισσότερες πληροφορίες. Όσον αφορά το τελικό καθεστώς, εκεί πέρα θα ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, γιατί εμεί έχουμε κάνουμε την ομαθητική πρόταση. Όσον αφορά όμω το περιεχόμενο, θα έχετε τι επόμενε ημέρε ένα έγγραφο με συγκεκριμένε πληροφορίε. Ένα άλλο στοιχείο είναι να αυξήσουμε την επίπτωση των ταμείων αυτών. Πώς το πετυχαίνουμε τώρα αυτό. Μέσω της θεματικής συγκέντρωσης έχουμε 11 θεματικούς στόχους που θα εφαρμόζονται και στα 5 ταμεία. Αναφερόμαστε κυρίως στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στο Ταμείο Συνοχής. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προτείνουμε μια θεματική συγκέντρωση που θα επικεντρωθεί σε ένα 80 60 ή 50% συγκέντρωση για τρεις συγκεκριμένου τομείς. Ε, έρευνα και ενημέρωση καινοτομία, ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οικονομία, οικονομική ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Το τελευταίο έχει αναφερθεί σε πάρα πολλές παρεμβάσεις σήμερα το πρωί. Ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Ακολουθούμε μια πολιτική που μέσα από την πάροδο των ετών έχει προσπαθήσει να κάνει ένα απολογισμό για το στόχους με τους οποίους, ε, τους οποίους χρησιμοδοτούμε μέσω των προγραμμάτων αυτών. Θέλουμε να αυξήσουμε περισσότερο την ορατότητα που δίνεται για τα αποτελέσματα αυτά. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε κοινού πλέον ε, δείκτες. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να δούμε καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πού χρησιμοποιούνται και γιατί χρησιμοποιούνται τα ταμεία αυτά. Όσον αφορά τώρα την εξάντε αιρεσιμότητα και πάλι εδώ πέρα θέλουμε εξ αρχή να υπάρχουν οι απαραίτητοι όροι οι οποίοι θα οδηγήσουν στην επιτυχία. Προτού χρηματοδοτήσουμε λοιπόν ένα ε, έργο, προτού δώσουμε χρήματα για την έρευνα, και τις μεταφορές, θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, να καταλαβαίνουμε πώς εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο στο γενικότερο σχέδιο που μπορεί να υπάρχει για την πόλη, για το κράτο μέλο και την περιφέρεια. Όσον αφορά επίσης τις επιδόσεις, θέλουμε ένα 5% της χρηματοδότησης να δοθεί βάσει του αν το πρόγραμμα πετυχαίνει αποτελέσματα. Όσον αφορά την μακροοικονομική αιρεσιμότητα, η συζήτηση αυτή ξέρετε ότι έχει σχέση όχι μόνο με την πολιτική συνοχής, αλλά έχει να κάνει και με τις γενικότερες πολιτικές οικονομικής διακυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την απλούστευση και αυτό αναφέρθηκε δύο-τρεις φορές. Ξέρετε ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τη δική μας πολιτική. Όλες οι πολιτικές χρηματοδότης στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου έχουν ως στόχο να πετύχουν και ένα συγκεκριμένο βαθμό απλούστευσης. Επομένως θα δείτε ότι τα πρώτα 80 άρθρα θα ισχύουν και και τα 5 ταμεία, που σημαίνει ότι οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να ανταποκριθούν σε πολλούς διαφορετικούς κανόνες. Έχουμε επίσης ε, πολλές διαφορετικές επιλογές όσον αφορά τη χρηματοδότηση από πολλά ταμεία και έχουμε και κάποιες νέες διατάξεις ε, προκειμένου να απλουστεύσουμε περισσότερο τα πράγματα. Τέλος, Προτού δώσω το λόγο στον αδελφό μου που θα μιλήσει πιο συγκεκριμένα για τι μεταφορέ. να σα πω ότι προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τι εταιρικέ σχέσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα και μα είχε πει ότι πρέπει να ενισχυθεί το μέσα αυτό στα μελλοντικά προγράμματα, μολονότι η πολιτική συνοχή ήταν ανέκαθεν μία από τι πολιτικέ η οποία είχε ως στόχο να φέρει κοντά και να προωθήσει τη συνεργασία πολλών εταίρων. Η εταιρική λοιπόν αυτή σχέση θα υπάρχει σε κάθε φάση του προγράμματος, δηλαδή και στην προετοιμασία, στην εφαρμογή και στην παρακολούθηση, αλλά θα υπάρχει και ένας κώδικας συμπεριφοράς που θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανταποκρινόμαστε ουσιαστικά στα αιτήματα της ΕΟΚΕ αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συγκεκριμένα της Επιτροπής σας. Στα πλαίσια του κοινού στρατηγικού πλαισίου ε, σας είπα ότι θα έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα σας δοθεί τις επόμενες εβδομάδες. Κατά αυτόν τον τρόπο όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομη. Μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στον συναδελφό μου που θα μιλήσει περισσότερο για τον ε, τομέα των μεταφορών. Um, ναι, ελπίζω όμω ο Μάικλ να μην μακρηγορεί στο τέλο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος ως προς τα θέματα μεταφορών. Αυτό που βλέπετε στον κανονισμό αντικατοπτρίζει τους άλλους κανονισμούς που διέπουν τις μεταφορές. Γι' αυτό μας ε, ε, απασχόλησε και η Λευκή Βίβλος ως προς τις μεταφορές και τα σύναφη. Οι κανονισμοί αυτοί που έχετε ενώπιόν σας αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για τις βιώσιμες μεταφορές. Τα βλέπετε στη θεματική και στις επενδύσεις. Επίσης προσπαθούμε να ε, υποστηρίξουμε τη, τις διατροπικές ε, βιώσιμες μεταφορές πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε και ανοιχνεύσαμε ορισμένους τρόπους μεταφορών και βλέπουμε και την εξάντε ερεσιμότητα η οποία βοηθάει τα κράτη-μέλη για να προωθήσουν ε, βιώσιμα σχέδια μεταφορών εγκαίρως και χωρίς προσκόμματα. Αυτό ακριβώς ε, προσπαθούν να καταφέρουν ε, όλα τα κράτη-μέλη στις διατροπικές. Αυτά τα ολίγα. Ο Μάικλ, για να συνοψίσει. <clears throat> Äh, ναι. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του συναδέλφου για την συνεισφορά τους και νομίζω θα συνεργαστούμε όπως είχαμε κάνει και με τη Λευκή Βίβλο για τι συγκοινωνίε. Θα γράψουμε ένα σχέδιο πριν παρουσιάσουμε την έκθεση 24 Απριλίου και μετά να ψηφίσουμε 31 Μαΐου. Οπότε 29 ή 30 Μαΐου θα έχουμε τη συζήτηση τη τελευταία. Δύο πράγματα ξέχασα. Πράξεις κάτι εξουσιοδότηση, δεν τις ανέφερα. Ο κύριος Ρικέ ήταν ο που ανέφερε. Και βεβαίως η Κομισιόν θα ήθελε για τα πάντα πράξεις κατεξιοδότηση για να ξεφορτωθεί και το Κοινοβούλιο. Αλλά πρέπει μετά να κατεβείτε στις ευρωεκλογέ. Αλλά για την ώρα εμείς είμαστε οι οπότε εγώ προσωπικά είμαι κατά του να σας δώσουμε ε, λευκή επιταγή. Θεωρώ ε, πως δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλιώς τι μας ψηφίζουν εμάς. Όχι θα μιλήσουμε κι εμείς. Και γι' αυτό και μιλάω για την ευρεία πλευσία του Κοινοβουλίου. Μάλιστα. Και κάτι ακόμα θέλω να αναφέρω. Κυρία Τικάου, πράγματι μπορεί να υπάρχουν ε, ανάγκες για δρόμους στα νέα κράτη-μέλη. Αλλά ξέρω πως κατά βάση επενδύουν στους δρόμους και παραμελούν τους σιδηροδρόμους. Αυτό ισχύει στη Ρουμανία. Ήθελα να ταξιδέψω με το τρένο, αλλά αναγκάστηκα δυστυχώς να πάω με το αυτοκίνητο. Ή μάλλον να με πάνε με σοφέρ, για να ακριβολογώ. Ε, για την ε, Ουγγαρία, την, την, την Πολωνία έχουν 1,2 ε, δις επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Και πρέπει να προσέξουμε, αν τα επόμενα έτη ολοκληρώσουμε ε, το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, τότε θα είναι πάρα πολύ αργή η σιδηρόδρομη γιατί θα έχει μετατοπιστεί όλη η κίνηση αλλού. Πρέπει να τα κάνουμε και τα δύο παράλληλα. Όπως μεταξύ Βερολίνου και Αμβούργου υπάρχουν σιδηρόδρομοι, παίζει μικρότερο ρόλο αυτοκινητόδρομος και σχεδόν καθόλου τα αεροπλάνο. Οπότε μπορούμε να έχουμε σιδηρόδρομους ε, που θα είναι και αρκετά αποδοτικοί. Δεν είμαι δογματικός και λέω όχι κανέναν ε, ούτε ένα νέο μέτρο δρόμου, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και το κλίμα και η κινητικότητα παίζει ρόλο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Μάικλ, ε, στις 31 Μαΐου θα ψηφίσουμε. Θα δούμε την έκθεση, την περιμένουμε και μετά θα ορίσουμε προθεσμία για τις τροπολογίες. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγουν οι πρωινές μας εργασίες. Θα επανέλθουμε στις 3 με την ε, παρουσίαση της μελέτης για το ΤΕΝΤΗ, για τα, τους ε, χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. Ευχαριστώ.